So, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me to open our today's Καλησπέρα. Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν δείτε το πρόγραμμά μας, στην μέση διάταξη, έχουμε μια μικρή αλλαγή. Άλλαξε η ημερήσια διάταξη, προτείνει το εξή. Το σημείο 12, ενεργός, ε, ενεργός διάλογος με τις πολίτες της Ευρώπης, θα εξεταστεί πριν από το σημείο 11 απαλλαγή του 2007, Τετάρτη πρωί. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται αυτή η αλλαγή, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις. Ως ήθιστε, θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων της 8ης Ιανουαρίου, 13ης Ιανουαρίου, Ακολουθούμε τη συνήθεια διαδικασία. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια που θα διαβιβαστούν προς τη γραμματεία μέχρι αύριο το πρωί, τα πρακτικά θεωρούν τους εγκεκριμένα. Πριν ξεκινήσουμε, να καλωσορίσουμε το νέο μέλος, το Πιέρ Μπριμπέτιτς, που κάθεται εκεί, αντικαθιστά, το Μισελ Ροκάρ. Κύριε Πριμπέτιτς, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πριν ξεκινήσουμε υπάρχει ένα σύντομο μήνυμα από την ομάδα μας του webstream της τοσελίδας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο σας, διαφορετικά θα εμφανίζεται στο διαδίκτυο λάθος όνομα, διότι όπως ξέρετε οι συνεδρία επιτροπής αυτής μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Με αυτή την ε, ανακοίνωση μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης η στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. Δίνω το λόγο στη Μαρία Ελένη Κοπά την συγκήτρια. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα σχέσεων με τη Βραζιλία και επομένως είναι αναγκαίο ένα συντονισμένο, συνεκτικό πλαίσιο για τη σχέση των δύο πλευρών. Θεωρώ ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων είναι προς το συμφέρον και των δύο και βασίζεται σε ιστορικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς δεσμούς, αλλά και στις κοινέ αξίες για δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Στην πρώτη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Ιούλιο του 2007, αποφασίστηκε από τις δύο πλευρές να εγκυνιαστεί μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση στη δεύτερη που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 2008, καθορίστηκε το πρόγραμμα δράσης. Στην έκθεσή μου έχω περιλάβει τα σημεία εκείνα που θεωρώ σημαντικά για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στα δύο μέρη, όπως πρώτον το γεγονός ότι η Βραζιλία είναι χώρα καθοριστικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ, δύο, ότι η Βραζιλία θα μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων στη Λατινική Αμερική, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης. Τρία, με δεδομένη την παγκόσμια οικονομική κρίση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία πρέπει να συνεργαστούν σε επίπεδο ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα. Και τέταρτον, όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η συμμετοχή της Βραζιλίας στα διεθνή φόρα μπορεί να συμβάλλει στην επανεξέταση του ρόλου των διεθνών οργανισμών κατά την εποπτεία και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και φυσικά μέσα η έκθεση περιλαμβάνει τα ζητήματα ενέργειας, βιοκαυσίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, μετανάστευσης, φτώχης κτλ. Στην έκθεση κατατέθηκαν 13 τροπολογίες. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι τις υπέβαλαν. Εξ αυτών οι έξι είναι μου και αφορούν την επικαιροποίηση της έκθεσης σε σχέση με τα αποτελέσματα της δεύτερης διάσκεψης που έγινε στο Ρίο το Δεκέμβρη του 2008. Τώρα, σχετικά με τις υπόλοιπες. Η τροπολογία 3 μπορεί να είναι αποδεκτή και είναι προσθέτει ένα στοιχείο το οποίο ε, νομίζω είναι σημαντικό. Η τροπολογία 4 μπορεί και αυτή να γίνει αποδεκτή. Η τροπολογία 6 ε, περιλαμβάνεται σε μια άλλη παράγραφο, την παράγραφο ε και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι και δεν, ε, την, ε, δεν είναι αποδεκτή. Η τροπολογία 7 ε, δεν μου είναι πολύ κατανοητή, γιατί έτσι κι αλλιώ οι αρχέ που αναφέρονται είναι οι προποθέσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό δεν είναι αποδεκτή. Ε, ε Επίσης πρόβλημα είχα και με την τροπολογία 8 όπου αναφέρει ότι η οικονομική κρίση πλήττει τα μειονεκτούντα άτομα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Η οικονομική κρίση πλήττει όλους οπότε δεν ε, μπορώ να τη δεχτώ. Η τροπολογία 10 ε, περιλαμβάνεται στην παράγραφο L Οπότε νομίζω ότι δεν προσθέτει κάτι. Και τέλος η τροπολογία 12 ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα και θεωρώ ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος ούτε το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής που είναι μια, ένα κείμενο γενικής στρατηγικής σε σχέση με τη Βραζιλία για να γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Ε, όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, έχω αποδεχθεί και έχω ενσωματώσει όσα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στη δική μου έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιο Ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Ο κ. Γιάννης. Έχετε το λόγο. Gracias, presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την εισηγητρία. που στην πρώτη έκθεση που ανέλαβε έχει κάνει μια αξιέπαινη εργασία και σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βασιλεία και την εμβάθυνση των σχέσεών τους. Είχα παρουσιάσει μια σειρά από τροπολογίες. Μία από αυτές έχει γίνει δεκτή η υπαριθμόν 3, τις άλλες η συγγήτρια δεν τις δέχτηκε. Μερικές γιατί μπορεί ήδη να περιλαμβάνονται στο κείμενο όπως η τροπολογία υπαριθμόν 6. Αλλά υπάρχει και μία άλλη, η 10. Αλλά δεν κατάλαβα εκεί το επιχείρημα βάσει του οποίου δεν θέλει να την συμπεριλάβει η συγγήτρια, γιατί αναφέρεται σε κάτι το οποίο δεν βρίσκεται μέσα στην έκθεση, έχει να κάνει με τη συνεργασία για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της διακίνησης των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας. Είναι <clears throat> ρήτρες που τις ε, ενσωματώνουμε εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, ιδίως με τρίτες χώρες <clears throat> της εμβέλειας της Βραζιλίας. Νομίζω ότι τα θέματα της διεθνούς τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της ε, λαθρεμπορίας ναρκωτικών είναι μια γενική και μόνιμη δυστυχώς απειλή για μας, για την ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια. Γι' αυτό πάντα σχεδόν αυτόματα εισάγουμε τα στοιχεία αυτά, τις μνήες αυτές σε μια έκθεση που αφορά συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δέχεται η τροπολογία 12 που έχει να κάνει με την ενίσχυση της συνεργασίας στην πυρηνική έρευνα. Το γνωστό σχέδιο ΙΤΕΡ, το πρόγραμμα θερμοπυρηνικής σύνδεξης σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία και γνωρίζουμε ότι στην ε, περίπτωση της παραγωγής ενέργειας από θερμοπυρηνική σύνδεξη αυτό δεν σημαίνει ότι φτιάνουμε ατομικούς σταθμούς, απλώς πρόκειται για μία έρευνα στην οποία αξίζει να υπάρχει συνεργασία στα θέματα αυτά. Και επίσης η Ελλάδα, η χώρα από την οποία προέρχεται η συγγήτρια, έχει συμμετάσχει σε πολλούς οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πυρηνική έρευνα, την θερμοπυρηνική σύνδεξη, οπότε πιστεύω θα ήταν εύλογο να υπάρχει και μια συνεργασία από την πλευρά της Βραζιλίας και μια ενσωμάτωση της Βραζιλίας στους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με έρευνα τέτοιου είδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος my plate. My plate. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κόπα για την εκθέση αυτή, η οποία έχει πολύ θετικές πτυχές σε σχέση με τη στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. Θέλω να την ευχαριστήσω που εδέχτηκε μια τροπολογία της δικής μου πολιτικής ομάδας σε σχέση με την ε, αναγνώριση του ηγετικού ρόλου που παίζει η Βραζιλία στη Λατινική Αμερική μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή αυτή. Είναι γεγονός ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους τρόπους, γίνεται με βάση την δημόσια παρέμβαση στην οικονομία, αντίθετα από αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν μπορέσουμε να έχουμε μια παρόμοια παρέμβαση δημόσια στην οικονομία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική καθώς και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντος μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι αναφέρεται η πολυμερή συνεργασία, τα διεθνή φόρου, φόρα, συνεργασία με τις ΗΠΑ, συνεργασία στα θέματα του περιβάλλοντος, αηφόρου αναπτύξεως, η αντιμετώπιση της μετανάστευσης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας των ΗΠΑ, ο ηγετικός ρόλος σε κοινωνικές πολιτικές της Βασιλείας, όπως παραδείγματος χάρη το η οικονομική προπολογισμική υποστήριξη προς αυτούς, νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια πολύ θετική προσέγγιση. Πέραν αυτής της τροπολογίας που έχει γίνει δεκτή, έχουμε και δύο ακόμα τροπολογίες στις οποίες εγώ θα ήθελα να επιμείνω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Η τροπολογία 7, η οποία αναφέρεται στο εξή ότι όταν μιλάμε για οικονομικές σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα, η οικονομική και εμπορική αυτή σχέση θα πρέπει να λάβει υπόψη την έλλειψη συμμετρίας που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι μια μόνιμη αίτηση της ομάδας μας να ληφθεί υπόψη η ασυμμετρία σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Βραζιλίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη πλευρά και επίσης υπάρχει τροπολογία 8 η οποία θεωρεί λέει η κυρία Κόπα ότι η κρίση θίγει όλους αλλά όχι όλους με τον ίδιο τρόπο πρέπει να επισημάνω. Επομένως και σε μια εταιρική σχέση μεταξύ ημών και της βασιλείας, μια στρατηγική εταιρική σχέση, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα απαραίτητα ώστε οι πιο αδύναμοι, οι λιγότερο προστατευμένοι να έχουν τη δυνατότητα να βγουν και αυτοί από την κρίση που δεν είναι αυτοί οι οποίοι τις δημιούργησαν, είναι η μεγάλη χρηματοοικονομική όμιλη σε παγκόσμιο επίπεδο που δημιούργησαν την κρίση και δεν έχουν καμία σχέση με τους εργαζόμενους ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα λιγότερο στη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ιάννα Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ελενκόπα για τη θαυμάσια έκθεση που μας υποβάλλει. Είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη σημασία στο να δώσει το Κοινοβούλιο μας μια άποψη και μια θέση να δώσει ως μέση στάση προς το Συμβούλιο σε σχέση με ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η εταιρική στρατηγικού χαρακτήρα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια μια χώρα κομβική, θεμελιώδης, όλο και πιο σημαντική στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Παίζει σημαντικό ρόλο λόγω και της πολιτικής και πολιτιστικής εμπειρίας που έχει αποκτήσει κυρίως με την ανάμειξη διαφόρων φυλών, λαών, ρευμάτων, πεπιθήσεων. που έχουν συνιστοσών, εν πάση που έχουμε διαφορετική ιστορική πορεία, όλο και περισσότερο αυτό είναι ένα σημαντικό παράδειγμα στον κόσμο στον οποίο ζούμε εγώ ως Πορτογαλέζα και ως σοσιαλίστρια. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη Βραζιλία, έχει πολλά να κερδίσει σε επίπεδο ποιότητος από τη σχέση αυτή με τη Βραζιλία μέσω ενό έντονου και στρατηγικού χαρακτήρα διαλόγου με τη Βασιλεία, μπορεί σε συντονισμό, σε συνεργασία με τη Βασιλεία στα Ηνωμένα Έθνη και στους χώρους πολυμερούς συνεργασίας να επιτύχει πάρα πολλά πράγματα και χάρη σε αυτήν τη συνέργεια προσπαθειών μπορούμε να είμαστε και οι δύο πλευρές αποτελεσματικοί. Εγώ συμφωνώ σχεδόν με όλες τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Νομίζω ότι οι, <clears throat> οι αντιρρήσεις που έθεσε ο Λουίς Γιάννης προηγουμένως σε σχέση με τη θέση της εισηγήτριας για τις μνήες του εμπορίου ναρκωτικών και της διεθνούς τροποκρατίας και τα λοιπά. Αυτά όμως ήδη περιλαμβάνονται στο κείμενο της έκθεσης. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια διαφορά απόψε μεταξύ του Λύς και της Ελένης για τα θέματα αυτά. Και εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε μια άλλη τροπολογία που προτάθηκε από τον Λουίς Γιάννης την 12 σε σχέση με τη συμμετοχή της Βασιλείας στο σχέδιο ΙΤΕΡ, θερμοπυρηνικής σύνδεξης. Την πρώτη φορά που είδα αυτή την ε, τροπολογία αντέδρασε όπως και η Ελένη. Αλλά κοιτάζοντα το θέμα αυτό περισσότερο, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η τροπολογία του κύριου Γιάννης είναι ορθή. Γιατί πράγματι στο πολυεθνικό αυτό σχέδιο το ΙΤΕΡ πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία. Και εμείς μιλάμε τώρα για την ανάπτυξη της ε, θερμοπυρηνικής σύνδεξης, όχι της ε, σχάσης που οδηγεί στην παραγωγή πυρηνικών βομβών. Η σύνδεξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική μέθοδος, η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου για την παραγωγή ενέργειας με τρόπο πιο καθαρό και πιο οικονομικά αποδοτικό από ότι η συμβατική πυρηνική σταθμή. Επομένως, νομίζω ότι έχει νόημα να συμπεριλάβουν και τη Βραζιλία σε αυτό το σχέδιο και επίσης, επειδή μας ενδιαφέρουν τα θέματα της μη διασποράς των πυρηνικών όπλων, Δεν θέλουμε λοιπόν οι επιστήμονες τη Βραζιλία ή τη Ινδία ή οποιοδήποτε άλλου κράτου να χρησιμοποιήσουν τι γνώσει για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, πυρηνικών οπλικών συστημάτων, είναι λογικό μέσα στα πλαίσια αυτά να μπορέσουμε να προσελκύσουμε την ε, Βραζιλία σε αυτό το σχέδιο, το οποίο οδηγεί σε μια καλύτερη άρθρωση σε επίπεδο εταίρων και καλύτερη συνεργασία για την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ. Mr. Rosing, please. Uh, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα μου, δανέζικα. Καλώς. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μεγάλος υποστηρικτής του προγράμματος ITER και παλιά έγινε μάχη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ιαπωνίας πάνω σε αυτό για το πού θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και οι Ιαπωνέζοι έδωσαν πάρα πολλά λεφτά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να πάει το πρόγραμμα στην Ιαπωνία. Όμως κατέληξε να είναι εν μέρη στη Γαλλία και εν μέρη στην Ισπανία. Η, ε, θα δημιουργηθεί βιομηχανία μέσω αυτού του προγράμματος η οποία βιομηχανία θα ασχοληθεί με, το, με τις νέες πηγές ενεργείας και είναι σημαντικό οι περισσότεροι δυνατοί εγκέφαλοι να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και οι περισσότερες χώρες στην προσπάθεια ανάπτυξη προγράμματο και θα πρέπει να αναπτυχθεί ο τομέα. Και όταν θα έχουμε μετακίνηση προ άλλε μορφές ενεργείας, τότε όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση τη ενέργεια. Αν θέλουμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα αυτό, στο ΙΤΕ δεν θα είναι δωρεάν, θα πρέπει να πληρώσουμε για να συμμετάσχουμε. Και λόγω των διαπραγματεύσεων και των μεγάλων ωφελιών που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες, και συμμετέχουσες βιομηχανίες. Λόγω όλων αυτών, προφανώς κάποιος πρέπει να πληρώσει για να συμμετάσχει. Άρα είναι σημαντικό να ανοίξουμε τις πόρτες για εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν. Θα είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσει το πρόγραμμα γρήγορα. Ίσως μετά από 50 χρόνια θα διατεθεί στο εμπόριο αυτή η ενέργεια, αλλά τώρα θα πρέπει να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρία Κοπάτο, για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Ε, ήθελα να πω πρώτον ε, στον κύριο ε, Γιάννη Μπαρνουέβο ότι ειδικά για το θέμα που αναφέρεται στην τροπολογία 10 υπάρχει, όπως ε, είπε και η Άννα Γκόμες, ακριβής παράγραφο που αναφέρεται συγκεκριμένα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρήματος, εμπόριο όπλων μικρού διαμετρήματος, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία. Άρα ε, η ε, τροπολογία αυτή σε κάθε περίπτωση είναι μια ε, επανάληψη. για το, τα θέματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Μέιερ Πλέτε και τον ευχαριστώ για την παρέμβασή του, είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τα μειονεκτούντα άτομα. Από την άλλη, επειδή έχει πάρα, πάρα πολύ, πολλές πλευρές αυτή η συζήτηση, δεν θα ήθελα να προσθέσουμε κάτι το οποίο αναφέρεται σε μία πλευρά μόνο των συνοπιών της κρίσης και γι' αυτό ήταν η δική μου αρνητική θέση σε αυτό. Τώρα για να ολοκληρώσω για το πρόγραμμα ITER για το οποίο τοποθετήθηκαν αρκετοί συνάδελφοι. Το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο όπως είπα γενικής στρατηγικής η παράγραφος στην οποία ο κύριος Γιαννιές Μπαρνουέβο ζητάει να γίνει αυτή η αναφορά στο πρόγραμμα ΙΤΕΡ είναι, μια γενική παράγραφος όπου αναφέρεται στην ανάγκη να αναπτυχθούν ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Όπως επίσης και η ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, συνολικά. Είναι λοιπόν μια γενική παράγραφος. Το να γίνει αναφορά σε ένα ειδικό θέμα, σε ένα ειδικό πρόγραμμα, όπως είναι το ΙΤΕ, χωρίς να γίνει αναφορά σε άλλα προγράμματα, σε άλλους τομείς, το θεωρώ ότι είναι μονομερές, θεωρώ ότι χάνει η παράγραφο στην ισορροπία της και επίσης εισάγει ένα θέμα το οποίο, για το οποίο δεν έχουμε κάνει επαρκή συζήτηση και είναι σχετικά αμφιλεγόμενο. Για το λόγο θα παραμείνω στη θέση μου σχετικά ε, με την παράγραφο αυτή. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για, την, ε, για τις παρεμβάσεις τους και ε, επίσης και την Επιτροπή αλλά και τη Γραμματεία για τη συνεργασία, ε, την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά την ε, σύνταξη του κειμένου. Και πάλι ευχαριστώ. you, Ευχαριστώ κύριε Κοπά. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα. Τώρα θα διακόψουμε για λίγο ένα αναμονή του, της άφεξης του πρόεδρου του Τατζικιστάν. Για λίγα λεπτά θα διακόψουμε. No, hammer. Uh, dear colleagues, uh, ladies. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Ραμόν, πρόεδρο της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, στην πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες και να καλωσορίσω και τα μέλη της αντιπροσωπείας του, ιδιαίτερα τον, ε, την Υπουργό Εξωτερικών κ. Ζαρίφη, τον, τους πρεσβευτές ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας ήρθατε με μεγάλη αντιπροσωπεία κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και τον κύριο Γιούστον επικεφαλής αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο Καζακστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. Ε, έχετε ξεκινήσει μια επίσημη επίσκεψη στο Βέλγιο με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, τον ε, Γενικό Γραμματέα κ. Σολάνα, τον Πρόεδρο Μπαρόζο, την κ. Φερο, Βάλνερ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Ντεχόπ Σέφερ και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κοινοβούλιο αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας μεταξύ των οποίων και για τη χώρα σας που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και ήταν ένα βασικό σημείο διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόσφατη στρατηγική της για την Κεντρική Ασία υπογράμμισε και το και το ενέκρινε αυτό και το κοινοβούλιο στο ψήφισμά του πριν από τον περασμένο Φεβρουάριο μετά το ψήφισμα ως Δεμήρ ότι δίνουμε μεγάλη σημασία για την σταθερότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κατσουδικαίου στην Κεντρική Ασία, ιδιαίτερα καθότι οι πολιτικές εξελίξεις ε, στην Κεντρική, στην Κεντρική Ασία και η σημασία της, κατά, της κατάστασης στη χώρα λόγω και της γενίας AIDS του Αφγανιστάν αυξάνουν την πολιτική και στρατηγική σημασία της. Στην πράξη, η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ Ένωση και Τατζικιστάν υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 4 και επικυρώνεται αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη. Δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από την Ελλάδα. Ενώ από πλευρά του το Τατζικιστάν το κύρωσε τη συμφωνία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο εισηγητή μα κύριο Πέτρελε θα εξετάσουμε τη συναφή την συμφωνία αυτή στο εγγύ μέλλον. Δεδομένη τη κατάσταση αυτή, θέλουμε να γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, την άποψή σα για τι εξελίξει στη χώρα αλλά και τι εξελίξει στην περιοχή σα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, που ήρθατε και σα δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα εξ αρχής να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη διαδικασία ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του Τατζικιστάς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς. Ιδίως κατά τα τελευταία έτη η διαδικασία αυτή εντάθηκε σημαντικά και ποιοτικά και ποσοτικά. Πιστεύω ότι η επίσκεψή μου αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μας και στο πολιτικό, οικονομικό, ανθρωπιστικό τομείς αλλά και στον τομέα της ασφάλειας και την ενίσχυση της, περιφερει... της συνεργασίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Θα ήθελα να πω ότι οι κοινοβουλευτικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τατζικιστάν ξεκίνησαν το 2004 και έχουν ήδη διεξαχθεί τρεις συναντήσεις ε, που συζήτησαν ζητήματα όπως την, το ρόλο του Κοινοβουλίου στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, την ενέργεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση ατόμων, τη διαφθορά και άλλους τομείς. Επιπλέον πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα ενίσχυσης των ε, περαιτέρω ενίσχυσης των διακοινοβουλευτικών δυνατοτήτων συνεργασίας. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων στο Ταντικιστάν, προσφέροντάς μας την πλούσια εμπειρία ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ανεξάρτητου ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να αναπτύξουμε και τις οικονομικές μας σχέσεις με την Ευρώπη. Διαπιστώσαμε ότι πέρυσι το εμπόριο σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τατζικιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήρθε σε 880 εκατομμύρια δολάρια, 20% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας. Οι σχέσεις αυξάνονται σημαντικά και τα τελευταία πέντε χρόνια τριπλασιάστηκαν οι εμπορικές μας ανταλλαγές. Προφανώς η οικονομική κρίση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ε, περαιτέρω σχέσεις μας. Η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές ιδιαίτερα λόγω της μείωσης ε, της ζήτησης πρώτων υλών, κυρίως ε, αλουμίνας και βάμβακος, έχει σημαντικές συνέπειες στην οικονομία. Ε, η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε σε μείωση κατά 50% της τιμής των προϊόντων αυτών και χρειάζεται να υπάρξει κοινή και ταχεία απάντηση στα προβλήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Ένα από τα μέτρα είναι η αύξηση των επενδύσεων από την Ευρώπη προς την οικονομία μας, που βρίσκεται σε ακόμα σε χαμηλότερο σχετικά επίπεδο. Το Τατζικιστάν έχει ε, υδροηλεκτρική δυνατότητα ενέργειας, αλλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ε, πολύ μικρό ποσοστό, μόνο 5%. Ωστόσο, η άρδευση, τα αρδευόμενα κομμάτια του, του Τατζικιστάν, παρά το ότι είναι ορεινή χώρα, δεν είναι πολύ μεγάλα, είναι λιγότερο από 1%. Χρειάζεται να αναπτύξουμε κατά συνέπεια την ηλεκτρική δύναμη για να βελτιώσουμε την οικονομία μας. Από αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε και να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού του Χόγκουν και να, κάτι που είχε ξεκινήσει κατά τη Σοβιετική περίοδο, διακόπηκε και ξαναρχίζει τώρα. Το, ο, υδρο, σταθμός αυτός του Ρόγκουν θα μπορούσε να σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, να λειτουργήσει εξαιρετικά θετικά όχι μόνο για μα, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή τη Κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένη και τη Ρωσία και του Ουσμπεκιστάν. Εξού και η σημασία σε περιφερειακό επίπεδο του υδροηλεκτρικού αυτού σταθμού. Οι συνέπειες, ε, ο, ο αυτός ο σταθμός θα βοηθήσει και την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνέπειων της αποξήρανσης της αράλης. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι γειτονικέ χώρες να μετάσχουν ε, άμεσα στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Ε, ε, είναι λυπηρό το ότι δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο η συνεργασία στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Επιπλέον, Επιπλέον, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξιακή πολιτική θα βοηθήσει την μείωση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας και την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων ε, διατροφής που έχουν τμήματα του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, μέσω του τάσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε σε μια σειρά έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και την οικοδόμηση νέων ε, οικονομικών δομών. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη βοήθειά σας. Ωστόσο, σήμερα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε πιο σημαντικές και πιο βαθιές διμερείς σχέσεις ε, για να υλοποιήσουμε την, ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κεντρική Ασία. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζεται σε ε, έμπιστους εταίρους στην Κεντρική Ασία. Η περιοχή μας αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις. Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές κοντά στα σύνορά μας θα επιτρέψουν να και στην Ευρώπη να, να, να βρεθεί σε καλύτερη θέση. Αυτό όμως απαιτεί χρηματοδότηση η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να στηριχτεί στην, ευρωπαϊκή, στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα, τον, το θρησκευτικό φανατισμό και, το, και την τρομοκρατία είναι ε, αναγκαιότητα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και, την, ε, συνέ, τις που θα έχει αυτό στην οικονομική αποκατάσταση του Αφγανιστάν. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας. Θα ήθελα να πω την άποψή μου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης συνόρων στο Τατζικιστάν. Κατά τα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 7.300.000 ευρώ για κατάρτιση ε, του προσωπικού στα σύνορά μας. Εμείς ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή της αυτή, αλλά κατά την άποψή μας τούτο δεν συγκρίνεται, τα ποσά δεν συγκρίνονται με την αναγκαιότητα επιτόπου. Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μεταξύ των άλλων χωρών της Κεντρικής Ασίας το Τατζικιστάν έχει το, μακρύτερο, το πιο μεγάλο το μήκο συνόρων με το Αφγανιστάν και άρα είναι το πιο ευάλωτο. Είναι λοιπόν έχουμε 1850 χιλιόμετρα σύνορα με το Αφγανιστάν και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια σύμφωνα με τις Ινωμένες με τα Ηνωμένα Έθνη, η βοήθεια στο Τατζικιστάν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της, ε, εμπορίας, του εμπορίου των ναρκωτικών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα από τα σημαντικά προβλήματα στο Τατζικιστάν σήμερα είναι η εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα, πρόοδος θα επιτευχθεί μόνο στις χώρες εκείνες που επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων. Οι νέοι Τατζίκοι θέλουν να ταξιδέψουν και να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο και περισσότεροι. Και πιστεύω ότι οι σπουδές των ανθρώπων αυτών στις χώρες της Ευρώπης θα ενισχύσει και τη φιλία μεταξύ των δύο, της χώρας μου και της Ευρώπης, αλλά θα ενσωματώσει στις, στις εθνικές παραδόσεις και αξίες την νέα ευρωπαϊκή διάσταση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα αυξήσετε την συμμετοχή των τατζίκων φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus Mundus και θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι δεν πληρούνται πλήρως οι προποθέσει του προγράμματος αυτού για το, για το Τατζικιστάν, αλλά θα έπρεπε να ενισχυθεί η δυνατότητα των νέων Τατζίκων να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στη Φρούντζε, όχι μόνο για τους Τατζίκους, αλλά για να προσελκύσουμε σπουδαστές από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, η αύξηση, η βελτίωση των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ Τατζικιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αξιών, των σχετικών αξιών και ελπίζω να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτό το μοναδικό και σημαντικό στόχο και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας επισημάνατε τις δυνατότητες που δίνονται για τη βελτίωση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τατζικιστάν. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και του εξειδικευμένου φορέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται με τις σχέσεις μας με την ε, ε, Κεντρική Ασία και χώρες όπως εσείς. Πρόκειται για την προσωπία η οποία ασχολείται με όλες τις χώρες στην περιοχή, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία. Και της αντιπροσωπείας αυτής προεδρεύει ο συνάδελφός μας, η συνάδελφός μας, η κυρία Γιουγκεβιτσιόνε, πρόεδρος ε, για την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και είναι και η πρώτη στην οποία θα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Καλωσορίστε για άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τιμή μου να σας βλέπω εδώ ως πρόεδρος της ε, Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας. Έχουμε ήδη δημιουργήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους εθνικούς σας βουλευτές. Έχουν γίνει κάποιες συνεδριάσεις και συζητήσεις, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα επικοδομητικές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κατέρωθεν. Δεν μπορώ παρά να δηλώσω λοιπόν ότι λυπούμε που η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασίας δεν έχει κυρωθεί ακόμα από ένα κράτος μέλος και θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την τυπική διαδικασία η οποία δεν μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις πλήρες δυνατότητες αυτού του πάρα πολύ πολύτιμου και πολύ χρήσιμου και για τις δύο πλευρές μέσω. Τον Οκτώβριο του 2007 έγινε μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Είχαμε ε, βουλευτές από τον Ντουσάμπε και φέτος έχουμε σχεδιάσει μια αποστολή στον Ντούσαμπε ευρωβουλευτών, την οποία περιμένω με ανυπομονησία. Θα ήθελα να τονίσω και πόσο σημαντική είναι η επίσκεψή σας εδώ, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη, Έχετε ήδη επισκεφθεί και μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λετωνία. Κάναμε μία σύντομη συζήτηση όταν φτάσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρω ότι θα επισκεφθείτε και άλλες δύο χώρες της Βαλτικής. Επισκεφθήκατε ήδη τη Λετωνία, θα μεταβείτε και στην Εστονία και στη Λιθουανία. Θα πάτε δηλαδή και στη χώρα μου. Κάναμε μία σύντομη συζήτηση με, τον, με την αυτοεξοχότητα, τον κύριο Πρόεδρο, για το σκοπό της επισκέψης τους σε αυτές τις τρεις χώρες της Βαλτικής. Θεωρώ ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες μεταξύ μας για τον δρόμο μας προς τον εκδημοκρατισμό, το δρόμο μας προς αξίες οι οποίες είναι ήδη ε, θεσπισμένες και καλά θεμελιωμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι στη διάρκεια της επίσκεψής σας στις χώρες αυτές θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε τα θέματα αυτά περαιτέρω. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μία ερώτηση την οποία ούτως ή άλλως έχω θέσει στον κύριο Πρόεδρο. Το Τατζικιστάν και ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει ίσως τον υψηλότερο αριθμό γεννήσεων στην περιοχή σε σχέση με άλλες ε, χώρες πλουσιότερες. Ίσως λοιπόν αν επισκεφτείτε τη Λιθουανία, τη χώρα μου, ο Πρόεδρος θα μπορούσε να μιλήσει λίγο για την ε, πείρα του και να μας πει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε εμείς την κατάσταση στη δική μου τη χώρα, διότι εμάς ε, η κατάστασή μας είναι η αντίστροφη ακριβώς. Έχουμε πτώση των γεννήσεων στη Λιθουανία και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Τέλος πάντων, για να σοβαρευτούμε, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πρόεδρο να μας πει κατά την άποψή του πόσο στενή μπορεί να είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ίσως και με τις χώρες της Βελτικής ε, πιο συγκεκριμένα. Προσωπικά διαπιστώνω ότι οι πάρα πολύ καλές ε, δυνατότητες που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνδράμει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στη βελτίωση των σχολείων και να διευκολύνει το νέο πληθυσμό του Τατζικιστάν να μορφωθεί. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2007 έως 2013 έχει εκταμιεύσει ένα κονδύλιο 250 εκατομμυρίων ευρώ για την ε, βοήθεια στις χώρες αυτές και πιστεύω ότι ένα πρόγραμμα όπως αυτό, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ε, είναι το μέλλον των χωρών αυτών. Είναι ένα πρόγραμμα για να δημιουργηθούν δημοκρατίες στις χώρες αυτές και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τις νέες κοινωνίες όπως αυτή του Τατζικιστάν. Σα καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω οι συνεδριάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να αποβούν χρήσιμε για εσά και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Ευχαριστούμε κυρία Γιουκεβιτσιόνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την πρώτη αυτή επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις που θα ήθελα να σας απευθύνω. Πρώτη, αναφερθήκατε στην, στον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι στο, έχει τη μέγιστη προτεραιότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβλέπετε κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, συγκεκριμένα προγράμματα, ούτω ώστε να συμβάλλει το Τατζικιστάν στην ε, ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεύτερο ερώτημα για το Αφγανιστάν. Αναφερθήκατε επίσης στο Αφγανιστάν. Παρακαλώ, κάντε μια αξιολόγηση της βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς αυτή τη χώρα. Της βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προς ε, αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ο Παλέτσκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you, Mr. President, for your... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις δηλώσεις σας και για την ετοιμότητά σας για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της χώρας σας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Περί συνεργασία συνεργασία είναι το ερώτημά μου. Όπως γνωρίζουμε είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας και των οικονομικών δεσμών. Ποιες είναι οι επιτυχίες περιφερειακής συνεργασίας? Συνεργασία μεταξύ Ταζικιστάν και γειτόνων της χώρας. Επίσης, τι γίνεται με τη σχέση μεταξύ Τατζικιστάν και χωρών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα <clears throat> θα σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει ο χώρος της Ευρώπης και των Βαλτικών χωρών και είναι η πρώτη μου επίσκεψη επίσημη ως Προέδρου του Τατζικιστάν στην περιοχή αυτή με στόχο να ενισχύσω τη συνεργασία και τους δεσμούς φιλίας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτύξουμε δεσμούς αμοιβαίας φιλίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των λαών των δύο πλευρών και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μέσα στις σημερινές συνθήκες χρειάζεται εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ημών και θέλουμε επίσης να θεσπίσουμε μια νομική βάση για τη συνεργασία μας, ένα νομικό πλαίσιο συνεργασίας για να υπάρξουν και περισσότερες επαφές σε επίπεδο προσώπων μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε όπως ελέγχθη προηγουμένως πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε υψηλό επίπεδο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι η επιθυμία μας να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η συνεργασία. Γιατί? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του κόσμου σήμερα και όπως ανέφερα προηγουμένως στην ε, παρουσίασή μου. Το Τατζικιστάν βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση, σε μια πολύ σημαντική γεωγραφική θέση, ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι. Έχουμε το πιο μακρύ σύνορο με το Αφγανιστάν, 1400 χιλιόμετρα. Και φυσικά δεν σας διαφεύγει η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στο Αφγανιστάν τα τελευταία 18-19 χρόνια μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης εξακολουθεί να υπάρχει μια κατάσταση αστάθειας στο Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν παίζει ένα κεντρικό ρόλο για την, για την εξασφάλιση της, ε, των συνόρων μεταξύ Τατζικιστάν και Αφγανιστάν και παίζει το ρόλο και ενός ενδιάμεσου χώρου ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να αποτραπεί η λαθρεμπορία όπλων και η διεθνή εγκληματικότητα και το λαθρεμπόριο όπλων. Γνωρίζετε όμως ότι το Τατζικιστάν αμέσως μετά την ανεξαρτησία του αντιμετώπισε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες ένα εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε σε υλικές ζημίες της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πολλές ανθρώπινες ζωής εμείς λοιπόν λέμε στο Τατζικιστάν, αν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου και εσύ κοιτάς από την άλλη πλευρά, δεν τον βοηθάς, οι φλόγες από το σπίτι του θα στραφούν και στο δικό σου σπίτι. Και το Τατζικιστάν είναι εν επιγνώση των προβλημάτων που προέκυψαν από τον πόλεμο και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Αφγανιστάν. Είχαμε και εμείς γνωρίσει την εμπειρία της τρομοκρατίας στο έδαφος μας. Έχουμε υποστεί και εμείς τις ε, καταστροφές που μπορεί να προκαλέσει ο, η Διεθνή τρομοκρατία. Γι' αυτό εγώ έχω κάνει μια έκκληση σε όλες τις χώρες να υπάρξει μια μια κατάσταση ασφαλείας με παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στα σύνορα Τατζικιστάν και Αφγανιστάν και εγώ ενοχλήθηκα με μια με μια διατύπωση που ακούστηκε εδώ ότι όλα αυτά είναι δικό σας πρόβλημα. Όχι, εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα αλλά ο κόσμος αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή είναι κάτι το οποίο το συμμεριζόμαστε όλοι. Είναι απαραίτητο να συνενώσουμε τις προσπάθειες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Το Τατζικιστάν είναι ενεργό εργό μέλος της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και συμμαχίας από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε. Ελπίζω λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο να αντιμετωπιστεί η διεθνής τρομοκρατία, η λαθρεμπορία ναρκωτικών και όπλων και μπορεί να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο στην περιοχή αυτή και σε αυτό περιλαμβάνουν και την επίλυση του προβλήματος του Αφγανιστάν. Το πρόβλημα λοιπόν του Αφγανιστάν Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να επιληθεί αυτό είναι οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Αυτή λοιπόν είναι η κύριη στόχη της παρουσίας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή της Βαλτικής. Ένα άλλο ερώτημα που ετέθη είναι πώς η δημοκρατία του Τατζικιστάν θα ενισχύσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της παιδείας. Όπως είπα προηγουμένως, το Τατζικιστάν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ενίσχυση των σχέσεων στον τομέα της παιδείας και θέλει να υποδεχθεί το παρακλάδι αυτό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Δημοκρατία στο έδαφος του, ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες όχι μόνο για τους φοιτητές από το Ταζικιστάν αλλά και για άλλους φοιτητές από την Κεντρική Ασία και το Αφγανιστάν, ώστε να μπορούν να έχουν μια παιδεία διεθνούς επίπεδου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα ήταν και μια σημαντική, μια ανεκτήμητη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση των ανθρώπων εδώ. Για τον ε, εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έληξε το 1997 με την Συμφωνία Συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο και επετέφθη η ειρήνευση μεταξύ μόνο και την, των ομάδων της αντιπολίτευσης. Μετά από αυτή την ειρήνη έχουμε καταφέρει σε πάρα πολλούς τομείς να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο και σήμερα υπάρχουν πολλοί φοιτητές και ιδρύματα ανώτερα της εκπαίδευσης στο Τατζικιστάν που βρίσκονται σε άνθηση. Είναι δεκάδες, δέκα φορές παραπάνω οι φοιτητέ. Υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στο Τατζικιστάν. Και γι' αυτό το λόγο ιδίω εμείς έχουμε ένα ταμείο, ένα προεδρικό ταμείο όπως λέγεται, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ταλαντούχους φοιτητές επί τη βάση της αξίας τους και της απόδοσής τους και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε περαιτέρω τα άτομα αυτά, να εκπαιδεύσουμε εμπειρογνώμονες και ειδικού για τους τομείς τους οποίους χρειάζεται το Τατζικιστάν. Ένα άλλο ερώτημα που ετέθη ήταν το συμφέρον του Τατζικιστάν σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πολλοί από τους Ευρωπαίους δεν ξέρουν καν που βρίσκεται το Τατζικιστάν. Αλλά το αλουμίνιο του Τατζικιστάν, ο χρυσός του Τατζικιστάν, εκ εξάγονται κυρίως προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα να προσελκύσουμε εταιρείε υψηλής τεχνολογίας, σύγχρονης τεχνολογίας από τις ευρωπαϊκές χώρες στο έδαφος μας, παραδείγματος χάριν το Τατζικιστάν μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν σχεδιάσει ένα διεθνές σχέδιο μεγάλης κλίμακος με ικανότητα παραγωγής 55.000 τόνων το χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν την παραγωγή επίσης και των πολιτήμων λίθων στο Τατζικιστάν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει τι ευρωπαϊκέ χώρε. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη συνεργασία σε οικονομικού τομεί, σε βιομηχανικού τομεί. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη μπορούν να προσφέρουν την σύγχρονη τεχνολογία του, κάτι το οποίο θα είναι συμπληρωματικό με του ε, πόρου που έχει τι πρώτε ύλε του Τατζικιστάν, συνδυάζοντα τα δύο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολύ σημαντικού στόχου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, προχωράμε σε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω σε εκείνους που σας, στα λόγια εκείνων που σας καλωσόρισαν. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τη χώρα σας. Έχω ένα ερώτημα όσον αφορά τα όσα είπατε αρχικά στην πρώτη σας παρέμβαση. Είπατε ότι μεταξύ χωρών της Κεντρικής Ασίας υπάρχει μια πολιτική μπλεμαργία αν θέλετε, πόθος για εξουσία. Θα ήθελα να επεκταθείτε όσον αφορά αυτή την έννοια. Τι εννοείτε με αυτή την πολιτική απληστία στην περιοχή. To switch to English, I can repeat this. Αν είναι πιο εύκολο μπορώ να σας απευθύνω την ερώτηση ξανά στα αγγλικά απάντηση. Μαχσουσαν, δαρμπορεί, Δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα για την ώρα και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε τον πρόεδρο. Διορθώθηκε το πρόβλημα. Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, θα ήθελα να πω, συνεχίζει ο πρόεδρος, θα ήθελα να πω ότι στην περιοχή εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και βεβαίως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας σήμερα είναι η χρήση της ενέργειας και η δάτινη πόρη. Η δάτινη πόρη της Κεντρικής Ασίας είναι μεγάλο θέμα. 60% των υδατίνων πόρων πηγάζουν από το Τατζικιστάν. Και χρησιμοποιεί μόλις το 5% των πόρων αυτών των υδάτινων Τατζικιστάν. Το υπόλοιπο 55% των υδατίνων πόρων της Κεντρικής Ασίας χρησιμοποιούνται από τις γειτονικέ χώρες. Και όπως προανέφερα, το Τατζικιστάν είναι ορεινή χώρα. 92% της χώρας μας αποτελείται από όρη και δεν έχουμε καλλιεργήσιμες γέες τόσες πολλές και ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως ε, χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά τη διοργάνωσή μας αυτούς τους τομείς να μπορέσουμε να συντάξουμε εκθέσεις βιωσιμότητας, να εφαρμόσουμε πιλωτικά προγράμματα, στατηγικά προγράμματα ε, στην περιοχή μας. Ε, Mr Zaleski. κύριος Ζαλέσκι έχει το λόγο. President, I'm here. Κύριε Πρόεδρε, The translation, all right? θα μιλήσω πολωνικά. Κύριε Πρόεδρε, όταν απαντήσατε στις ερωτήσεις των συναδελφών, αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και εμένα ιδιαίτερα, το θέμα της παιδείας. Όταν μιλάμε για το μέλλον και το νέο πληθυσμό σας, θα ήθελα να σας πω ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ ακριβή μένα, αλλά αργότερα αποφέρει καρπούς. Και παρά το γεγονός ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να υπάρχουν ανταλλαγές ε, μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας σας, ε, θα πρέπει να μας πείτε και τι έχετε να προσφέρετε εσείς στο Ταζικιστάν. Θα καλοδεχτείτε Ευρωπαίους ερευνητές που θα έρθουν στη χώρα σας και θα μπορέσουν να βοηθήσουν και την ίδια σας τη χώρα προγράμματα, για παράδειγμα, εργοστασίων υδροελεκτρικής ενέργειας ε, ή κάποια άλλα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να ε, διεξαχθούν σε πιο ανθρωποκεντρικά θέματα επιστημονικά. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πρώτο και πολύ καλό βήμα για να υπάρχουν καλές ε, σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της πρωτεύουσα μου είναι εδώ σήμερα και συνεργάζεται, υπέγραψε σήμερα μία συμφωνία με τα βελγικά πανεπιστήμια για ανταλλαγή και φοιτητών και διδασκόντων. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων του Βελγίου και του Τατζικιστάν και βεβαίως θέλουμε να καλέσουμε τους ε, ερευνητές σας. Υπάρχουν τομείς ε, πολλοί που μπορούμε να συνεργαστούμε. Σήμερα οι ε, φοιτητέ από 24 χώρες του κόσμου παρακολουθούν μαθήματα στο, στα πανεπιστήμια μας. Δεν είναι και κακό το ποσοστό. Χρειαζόμαστε να μας βοηθήσετε, χρειαζόμαστε τους εκπαιδευτικούς σας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ειδική στον τραπεζικό τομέα και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχουμε μία πρεσβεία εδώ, μία πρεσβεία στη Βρετανία, στη Γαλλία άλλη πρεσβεία και μια ισχυρή και δραστήρια συνεργασία με τις χώρες αυτές. Στο Βέλγιο ξεκινάμε τώρα την συνεργασία μας. Ε, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι σε εμά και μπορείτε να έρθετε και εύκολα γιατί παίρνετε τη βίζα κατευθείαν στο αεροδρόμιο στο Ντουσάμπε. Η κυρία Ντεκέιζερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα από πλευράς της ομάδας μου να σας καλωσορίσω και να πω ότι για πολλούς από εμά, πολλοί από εμά δια... ανακαλύπτουμε τη χώρα σας που δεν την ξέραμε. Στην παρέμβασή σας μιλήσετε για δύο θέματα που ως γείτον χώρα του Αφγανιστάν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Είπατε ότι ήσασταν δραστήριοι στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και αναφέρετε ότι η εταιρική σας σχέση με την Ευρώπη αφορούσε και την καταπολέμηση της, του λαθεμπόριου όπλων. Το ερώτημα μου είναι απλό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως συγκεκριμένα πώς αντιμετωπίζετε τα δύο αυτά ζητήματα. Λαθεμπόριο όπλων και λαθεμπόριων ναρκωτικών στη χώρα σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε ότι δεν ξέρετε το Τατζικιστάν. Η πρωτεύουσά μας η Ντουσάμπε είναι μια πόλη στην οποία η μόνη στρατιωτική, ξένη στρατιωτική δύναμη που βρίσκεται εκεί είναι η γαλλική. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Γαλλία. Βλέπετε ότι μερικές φορές συνεργαζόμαστε με τον γαλλικό στρατό που χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο μας. Ε, οι Γάλλοι έρχονται, υπέβαλαν αίτημα, δεν θέσαμε όρους, δεν το διαπραγματευθήκανε. Μόλις πήρα την επιστολή που μου ζητούσαν βοήθεια, τους έδωσα την άδεια αμέσως Διότι μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλους η σταθερότητα στην περιοχή, στο Αφγανιστάν ιδιαίτερα. Θέλουμε να έχουμε έναν γείτονα ειρηνικό για τη μάχη κατά των ναρκωτικών. Μέχρι το 1996 δεν είχαμε ούτε μία περίπτωση κατάσχεσης ηρωίνης στη χώρα μας. Μετά το 96 απογοητευτήκαμε, γι' αυτό ζητήσαμε την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. και των διεθνών οργανισμών. Συστήσαμε μια υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών, η υπηρεσία αυτή υπάρχει εδώ και 7 χρόνια και δουλεύει στο Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν. Έχουμε ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την καταστροφή εργαστηρίων κάνουμε κατασχέσεις 40 με 50 τόνων ναρκωτικών τον χρόνο. Εσείς στην Ευρώπη πόση ηρωίνη κατάσχετε. αν δεν τα συγκρίνετε και σε σχέση με, και με τα ποσά που δαπανούν οι μεν και οι δε για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει να έρθετε να μας βοηθήσετε να χτυπήσουμε το εμπόριο ναρκωτικών σε εμά από το να περιμένετε να φτάσουν τα ναρκωτικά σε εσά. Η χώρα μας είναι μια χώρα που αποτελεί το μαξιλαράκι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ Αφγανιστάν και Ευρώπης. Ασία είναι και, ε, και η χώρα μας, αλλά ε, δυστυχώς σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει συμφωνία για το τι είναι ναρκωτικό και πώς καταπολεμάται το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ε, ο κύκλος εργασιών που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο. Ιδίως δε, μετά την το ξεκίνημα της αντιτρομοκρατικής ε, μάχης στο Αφγανιστάν τετραπλασιάστηκε η παραγωγή ε, ναρκωτικών στο Αφγανιστάν και πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μου δεν καταναλώνονται ναρκωτικά, δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, εξάγονται όλα. Η ρίζα του κακού δεν είναι στη χώρα μας. Κύριε Ντεκεζέρ και πάλι, απλώς θα ήθελα να πω στον κύριο ότι είμαι Βελγίδα, όχι Γαλλίδα. Euh, uh, ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι Αμερικάνο, είμαι Βρετανό, λέει ο κύριο Τάνοκ. Ούτε Ιρλανδό δεν είμαι. Ένα τέταρτο Ιρλανδό το πολύ. Πρόσφατα το Κυργιζιστάν έκλεισε τη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί πριν από 10 μέρε και μετά από λίγε μέρε πήρα ένα μεγάλο δάνειο από τη, από τη Ρωσία. Βλέπετε αυτό να είναι μια ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή σα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τη ISAF στο Αφγανιστάν όπου υπάρχει μια ε, μεγάλη, μια παραδοσιακή μειονότητα των Τατζίκων που είναι εχθροί των Ταλιμπάν. Παραδοσιακά είπατε ότι τη δεκαετία του 90 υπήρξε ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Ισλαμιστών και πιο κοσμικών δυνάμεων. Επελήφθη το πρόβλημα αυτό και θέλω να σα συγχαρώ. Αλλά ποια είναι τα θετικά διδάγματα που μπορούμε να πάμε στη Δύση από το παράδειγμά σας και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Παλαιστινιακά εδάφη όπου υπάρχει η κοσμική Φατάχ και η Ισλαμιστική Χαμά. Κάτι το οποίο ε, φάνηκε και με την τρομερή αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να μάθουμε κάτι από τη δική σας εμπειρία για να μπορέσουμε μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο να ξεπεράσουμε αυτές τις διαιρέσεις και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι και οι σχέσεις σας με τους Ιρανούς ομοεθνείς σας κατά κάποιο τρόπο που είναι συγγενείς σας ως λαός και την προσπάθεια του πρόεδρου Ομπάμα να επιλύσει την αντιπαράθεση με το Ιράν και να το πείσει να σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ. Για την βάση στο Μανάς μπορείτε να ρωτήσετε τον πρόεδρο του, του οι βάσει του Τατζικιστάν είναι ανοιχτέ για όλες τις δυνάμεις της ΙΣΑΦ και τη διεθνή δύναμη στο Αφγανιστάν. Και το Τατζικιστάν έχει εκφράσει την απόλυτη διαθεσιμότητά του να δώσει διευκολύνσεις για την ΑΙΣΑΦ σε ό,τι αφορά εγκατάσταση στρατευμάτων και επικοινωνίε και τέτοια συναφή ζητήματα. Το θέμα της βάσης του Μανάς είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο μπορεί να δώσει απάντηση μονάχα ο, το Κυρκυζιστάν. Μόνο μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να επιληθεί το θέμα αυτό. Και σε ό,τι αφορά βέβαια το παράδειγμα αυτό που αναφέρατε για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και αυτοί μπορούν να επιλύσουν μόνο τους. Για τον εμφύλιο πόλεμο στο Τατζικιστάν, το Τατζικιστάν έχει υποστεί μια τεράστια τραγωδία μέσα σε ένα και μόνο χρόνο δύο πέντε πρωθυπουργοί και δύο πρόεδροι παρετήθηκαν και αντιμετωπίσαμε μία μεγάλη παρέμβαση από εξωτερικές ομάδες και υπήρξαν και ορισμένες ομάδες οι οποίες θέλανε να αλλάξουν το θεσμικό ιστό της χώρας μας. Το θεσμό της Προεδρίας του Τατζικιστάν. Ευτυχώς καταφέραμε να υπερνικήσουμε αυτό το πρόβλημα. Κάναμε οκτώ γύρους διαπραγματεύσεων για να επιτύχουμε την ειρήνευση και μαζί με την ομάδα της Ενωμένης Αντιπολίτευσης στο Τατζικιστάν και με την αρρωγή φορέων από τη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι διαπραγματεύσει είναι ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου. Δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί η ειρήνευση και η σταθερότητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να επιτύχουμε να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από ένα τραπέζι και να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμφιλίωσης και συνεννόησης. Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς όλα τα λεπτομεριακά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εμπειρία που έχουμε καταγάγει στο Τατζικιστάν για την επίτευξη της ειρήνης. Δεν μπορώ σε μία ή δύο ώρες να τα περιγράψω όλα αυτά τα στοιχεία. Τα Ηνωμένα Έθνη, η προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. οι σχέσεις μας με χώρες όπως είναι το Ιράν, μπορώ να πω ότι από πολιτιστική και ιστορική άποψη είμαστε πολύ κοντά στο Ιράν. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Και θέλω να πω, όπως ε, είπα προηγουμένως, να επαναλάβω, ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει να λυθούν τα προβλήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να υπάρξουν οι ειρηνικέ διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θέσουν επιτάπητος όλα τα εκρεμή θέματα για να μπορέσουν να επιληθούν. Δεν μπορούν να υπάρξουν στρατιωτικές λύσεις για τις διαφορές αυτού του είδους. Το Ιράν δεν είναι το Αφγανιστάν, ούτε το Ιράκ. όλες οι επιθέσεις που έχουν γίνει σε στρατηγικό επίπεδο πλήττουν κυρίως τον άμαχο πληθυσμό. Και επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι η Ιρανική πλευρά έχει δείξει την πρόθεσή της και τη διάθεσή της να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στον πολιτικό χώρο. πρέπει το Ιράν να αντιμετωπιστεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Αν σήμερα λοιπόν το Ιράν ακολουθήσει μια διαδικασία ανάπτυξης ενός πυρηνικού προγράμματος, θα πρέπει να το αφήσουμε να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία και να γίνει αυτό μέσα στα πλαίσια μιας στενής συνεργασίας με τους διεθνείς φορείς στο τομέα της ενέργειας είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει αντιμετώπιση αυτού του προγράμματος, να υπάρξει ειρηνική διαπραγμάτευση. Οι Ιρανοί έχουν μια βαθιά και μακραίωνα ιστορία προέρχονται από τον περσικό πολιτισμό και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν ειρηνικά να διαπραγματευτούν και να επιλύσουν όλες τις διαφορές τους με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτά θα ήθελα να σας πω. Thank you. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μία ακόμα ερώτηση για το Αφγανιστάν. Διότι γίνεται μια αναθεώρηση στι ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Θα ήθελα να ξέρω τι συμβουλή θα δίνετε εσεί στη νέα Αμερικανική κυβέρνηση, σε εμά στην Ευρώπη. Τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να αυξήσουμε τη στρατιωτική μα παρουσία ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο διπλωματία. Θα πρέπει να μιλήσουμε με του Ταλιμπάν ή κάποιο κλάδο τέλο πάντων των Ταλιμπάν ε, τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να γίνει βάσει της γνώσης σας ε, για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, σε όλες μου τις δηλώσεις, ε, σε όλες μου τις ομιλίες και συνεδριάσεις που κάνω στο Διεθνή Στίβο, χρησιμοποιώ την προσωπική μου άποψη για το Αφγανιστάν. Ξέρουμε ότι έχουμε πολιτικές εκλογές, ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός στο Αφγανιστάν, θα έχουμε εκλογή Προέδρου και πρόκειται για μια πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή για, την, για το Αφγανιστάν. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά. προκειμένου να προλάβει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκύψει από παράνομες ομάδες. Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη πολιτική κατάσταση. Το Αφγανιστάν θα πρέπει να διατηρήσει πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας με όλους τους ε, φορείς, τους οργανισμούς ε, του Αφγανιστάν και θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλους τους ε, παράγοντες ε, και τις ε, διάφορες εθνότητες και εδώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε όλες μας τις δυνατότητες. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να κλιμακωθεί η κατάσταση με τις ομάδες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διότι αυτό θα αποτελέσει απειλή για όλη την Κεντρική Ασία. Όσον αφορά την προετοιμασία των πολιτικών εκλογών στο Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν εξέφρασε την ετοιμότητά του για την ε, παροχή αρρωγής ε, σε όλους τους τομείς, καθώς επίσης και το γεγονός ότι είναι διατεθειμένο να βοηθήσει τους Αφγανούς να φύγουν από την ε, παραγωγή και καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών και να περάσουν στην παραγωγή άλλων ε, προϊόντων ώστε να περάσουν στην νομιμότητα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε έτσι να λύσουμε σε κάποιο βαθμό και το θέμα της παράνομης των ναρκωτικών. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο για την ενίσχυση των ε, ε, υπηρεσιών ασφαλείας του Αφγανιστάν. Η ανθρώπινη ενότητα βέβαια των χωρών που υποσχέθηκαν να βοηθήσουν και να συνδράμουν το Αφγανιστάν ε, στην ανοικοδόμηση των αστυνομικών αρχών του και των αρχών ασφαλείας δεν βοήθησε όσο είχε πει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορέσετε να μας πείτε λίγα λόγια για τις ε, τωρινές και τις μελλοντικές ε, σχέσεις της χώρας σας ε, στον επιστημονικό τομέα. Πριν από μερικά λεπτά, νομίζω ότι απάντησα ήδη στο ερώτημα αυτό. Βεβαίως, Υποστηρίζουμε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα το Τατζικιστάν, βλέπετε, χρειάζεται την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και χρειαζόμαστε στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα αυτό. Αν επί σήμερα τα προγράμματα τα υδροελεκτρικά έχουν στατική σημασία στο Τατζικιστάν χωρίς υψηλή τεχνολογία θα ήταν αδύνατον επιτυχώς να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό βλέπετε χρειαζόμαστε την υψηλή τεχνολογία. Επισκέφτηκα ευρωπαϊκές χώρες, ήρθα στις Βρυξέλλες και χαίρομαι, είμαι ικανοποιημένος που είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ μαζί σας και σας προσκαλώ έτσι ειλικρινά να έθετε να επισκεφτείτε επίσημα το Τατζικιστάν. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα της χώρας μας για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα το Τατζικιστάν και να έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε τη στέγη του κόσμου που είναι ένα κομμάτι του Τατζικιστάν. Σα Все. Большое спасибо. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτησή μας, για τη χρησιμότατη παρουσίασή σας, τις συμβουλές, τα σχόλια σχετικά με προβλήματα της πολιτικής Πασκή Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Θα ήθελα να πω στη γλώσσα σας ότι σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. finally. So, colleagues, let's start with our next item. Ας αρχίσουμε το επόμενο θέμα μας, αγαπητοί συνάδελφοι, ανταλλαγή απόψεων με τον καθηγητή Φάουστο Ποτσάρτ, ε, φέτη στο Διεθνή Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία στη Χάγη. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω κύριε καθηγητά υπήρξε δικαστής στο δικαστήριο από το Φεβρουάριο του 2000 αρχικά ξεκίνησε στο κυρίως δικαστήριο μετά πήγε στο εφετείο είναι και δικαστής στο εφετείο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα και ήταν και πρόεδρος του δικαστηρίου από τον Νοέμβριο 2005 μέχρι πέρσι. Ο καθηγητής, καθηγητέ Ποκτσάρ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχετε περίπου 15 λεπτά να προβείτε στην αρχική σας παρουσίαση και μετά θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων, μάλλον ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση συνεδρίαση. Όπως ξέρετε από το περασμένο Νοέμβριο δεν είμαι πλέον πρόεδρος ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Έχει εκλεγεί πρόεδρος ο συνάδελφος ο Πάτρικ Ρόμπινσον και παρά το γεγονός ότι θα ήθελε να έρθει αυτοπροσώπος να σας μιλήσει, δυστυχώς προεδρεύει ακόμα μια δίκης η οποία απαιτεί ε, καθημερινά εισακροάσεις θα έρθει βέβαια με τα χαράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον όταν θα του επιτρέψουν υποχρεώσεις του να έρθει. Θα σας μιλήσω σήμερα ως εφέτης ε, του δικαστηρίου κατόπιν εξουσιοδότησης του Πρόεδρου και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτό το πάρα πολύ πελίτιμο φόρουμ και να σας ε, παρουσιάσω και κάποιες ιδέες για την ε, παρουσία μου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σας δώσω καταρχάς κάποια στοιχεία. Σε μία δεκαετία ύπαρξης του δικαστηρίου, από τότε δηλαδή που συστάθηκε το 1993, έχουμε παραπέμψει 161 άτομα και μόνο δύο είναι ακόμα ελεύθερα. Σήμερα Έχουμε διαδικασίες ε, κατά 116 ατόμων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχουν και κάποιες ε, ανοιχτές ε, υποθέσεις ακόμα για 45 άτομα, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται ακόμα ήδη στη διαδικασία της έφεσης. Όπως έχω πει επανειλημμένως όταν ήμουν πρόεδρος του δικαστηρίου, το δικαστήριο είχε ως στόχο να συνεισφέρει στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες που είναι απαραίτητος για την ε, αποκατάσταση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην ε, περιοχή, αλλά να μην είναι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην περιοχή. Πρόκειται για ένα καθήκον στο οποίο ένα δικαστικό ίδρυμα δεν είναι ίσως ο πιο αρμόδιος φορέας. Είναι βέβαια κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να συνεισφέρει σε κάποιο βαθμό σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα που αφορούν την ε, λεγόμενη στρατηγική ολοκλήρωση, completion strategy του δικαστηρίου. Η στρατηγική αυτή ε, ξεκίνησε από το ίδιο το δικαστήριο στις αρχές της δεκαετίας και υποστηρίχθηκε και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητές μας και να παραπέμψουμε τις υποθέσεις ε, στα δικαστήρια της πρώην Ιουκοσλαβίας μόλις τα δικαστήρια θα είναι πρόθυμα και σε θέση να κάνουν τις ε, ε, δίκες εκεί. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει ασχοληθεί με πολύ περιορισμένο αριθμό υποθέσεων. Μιλάμε για 161 υποθέσεις, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την περιοχή Αναφέρονται σε χιλιάδες υπετίους οι οποίοι έχουν προσαχθεί στο δικαστήριο. Τα στοιχεία βέβαια δεν είναι επίσημα, αλλά υπάρχουν ε, στρατηγικές και στην περιοχή για την αντιμετώπιση των υποθέσεων αυτών. Πώς ε, προσπαθήσαμε να παραπέμψουμε αυτές τις υποθέσεις ε, στις περιοχές. Καταρχάς, παραπέμποντάς τους κάποιες υποθέσεις που είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στο δικαστήριο. Είχαμε περίπου 14 άτομα τα οποία τα στείλαμε πίσω στην περιοχή τους Τις περισσότερες ε, στο δικαστήριο στη Βοσνία Ζεγοβίνη έχουμε στείλει και δύο υποθέσεις στην Κροατία και μία στην Σερβία. Τα άτομα αυτά λοιπόν είναι υπόδικα στις χώρες τους. Και προς το παρόν είμαστε ικανοποιημένοι διότι τα εγχώρια δικαστήρια αντιμετωπίζουν αυτές τις υποθέσεις με δίκαιο τρόπο όπως αναγνωρίζει η έκθεση του ΑΣΕ αλλά και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επίσης, έχουμε μεταβιβάσει και ανακριτικό υλικό στο, στα δικαστήρια των περιοχών για περιπτώσεις σε οποίες δεν υπήρχε προσαγωγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά ήταν στη φάση της ανάκρισης και της έρευνας. Αυτό το υλικό απεστάλλει λοιπόν στις περιοχές προκειμένου οι εισαγγελικέ αρχές ε, των χωρών αυτών να ασχοληθούν με τις υποθέσεις αυτές. Ένα τρίτο μέτρο ήταν να βοηθήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ε, περιοχή δίνοντας ε, δηλώσεις, στοιχεία, υλικό καθώς επίσης και συνεντεύξεις για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ώστε να γνωστοποιηθεί το έργο του δικαστηρίου και να εποφοληθεί από αυτή την εμπειρία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το εθνικό ποινικό σύστημα, το τοπικό ποινικό σύστημα ε, όταν θα αντιμετωπίσει αυτές τις υποθέσεις. Εξετάζοντας λοιπόν αυτή τη ε, στρατηγική ολοκλήρωση στο σύνολό της, θεωρώ ότι πρόκειται για μια στρατηγική η οποία έχει εκπονηθεί όχι μόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δικαστηρίου, αλλά και για να ευνοηθεί η συνέχεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων για τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις χώριες αρχές προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να επιστραφούν αν θέλετε οι, οποίες, ε, ε, οι δραστηριότητες αυτές οι οποίες ξεκίνησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ακριβώς γιατί τα τοπικά δικαστήρια δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις υποθέσεις. Υπό αυτή την ε, οπτική γωνία πρόσφατα υιοθετήσαμε μια σειρά από μέτρα καθώς επίσης και μια μορφή συνεργασία η οποία δεν υπήρχε στον αρχικό κανονισμό. Ε, έχουμε δηλαδή τοπική συνεργασία ε, υπό την έννοια ότι ένα τοπικό δικαστήριο θα πρέπει να συνεργάζεται με το ποινικό δικαστήριο, ώστε εμείς ως Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές και συστήσαμε μια διαδικασία μέσω της οποίας ε, τα τοπικά δικαστήρια ή οι συμμετέχοντες στα τοπικά δικαστήρια να μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικό υλικό, σε έγγραφα ε, τα οποία ε, διαθέτει το δικαστήριο και από εκεί και πέρα θα εξετάζεται ε, από το δικαστήριο η διάθεση αυτού του εμπιστευτικού υλικού, λαμβάνοντας φυσικά όλα και τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, όπως επίσης το θέμα της προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων. Για τον ίδιο λόγο και προκειμένου τα τοπικά δικαστήρια να μπορέσουν να εργαστούν καλύτερα και να είναι σε θέση να κατανοήσουν και πολύ καλύτερα τι κάναμε εμείς, Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια κάποια μορφή εταιρική σχέση μεταξύ των δικαστηριών αυτών, όχι μόνο ε, συνεργασία του μακρόθεν, αλλά και με συνεδριάσεις κοινέ, με συζητήσεις. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που αφορά στις ε, δράφορες δραστηριότητε του, να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα μέσω συζήτησης με τους τοπικούς δικαστές και τους δικαστές ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις ε, διαδικασίες του δικαστηρίου και στην ομολογία, ε, δημιουργήθηκαν δύο μνημόνια συνεννόηθης, ένα με τη UNICRI που είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την ε, καταπολέμηση του εγκλήματος και η έδρα του βρίσκεται στο Τωρίνο και με την ODIR που είναι ένας οργανισμός στο ΑΣΕ Uh, για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να μπορέσουμε ε, να δούμε και τι ακριβώς γίνεται σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Ετοιμάσαμε ένα έγγραφο το οποίο ε, παρουσιάζει τα όσα έκαναν οι δικαστές ε, για τα ε, εγκλήματα κατά ε, τη ανθρωπότητα και τα εγκλήματα πολέμου. Αυτό το εγχειρίδιο έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί και τη βάση συζήτηση για το πώς ε, τα διεθνή δικαστήρια ή τοπικά δικαστήρια όπως το δικαστήριο στο Σαράγεβο και ε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει μετά από αυτό το πρώτο πείραμα που είχαμε στο διεθνή δικαιοσύνη δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες υποθέσεις ε, να τις παραπέμψουμε στα τοπικά δικαστήρια, αλλά θέλουμε να έχουμε μια βάση ώστε τα όσα θα γίνουν στα τοπικά δικαστήρια να είναι μια συνέχεια αυτών που κάνουμε εμείς σε διεθνές επίπεδο. Ε, και οι δύο οργανισμοί και ο Γιούνικρη και ο Ντύρ δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν για την ε, μεταβίβαση αυτών των πρακτικών στα τοπικά δικαστήρια και εμείς προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει μία πτυχή την οποία επεξεργαζόμαστε επί του παρόντος και δεν έχει απόλυτη σχέση με την ε, απόδοση δικαιοσύνης. Θα θέλαμε οι δραστηριότητες του δικαστηρίου να γνωστοποιηθούν στο κοινό στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παρά το γεγονός ότι κάναμε προσπάθειες προσέγγισης, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι απλοί πολίτες να κατανοήσουν τι ακριβώς κάνουν τα διεθνή δικαστήριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τους νομικούς ε, σε κάποιες περιπτώσεις να διαβάσουν μία απόφαση δικαστηρίου, μία απόφαση ενός διεθνούς δικαστηρίου. Μία ιδέα λοιπόν που είχα κάποια στιγμή και προσπάθησα να μοιραστώ με τους υπολείπους, κυρίως στη Βοσνία, ήταν να υπάρχουν κάποια κέντρα ε, ως μνημεία όπου θα μπορούμε να εξηγούμε στους απλούς πολίτες, στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό, πώς συνέβησαν αυτά τα πράγματα και πώς λειτουργεί η διεθνής δικαιοσύνη και φυσικά από εκεί και πέρα θα υπάρχει πλήρης ε, πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα ε, και τα κέντρα θα έχουν πρόσβαση στο υλικό του δικαστηρίου. Τα περισσότερα βέβαια από αυτά βρίσκονται ήδη στο διαδίκτυο και το πρόβλημα είναι ότι η τεχνική πρόσβαση δεν είναι επαρκής ώστε να γνωστοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία στο ευρύ Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το τι θα κάνουμε όταν θα κλείσει το δικαστήριο. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούν να κλείσουν με το πέρας της εντολής του Διεθνούς Δικαστηρίου για την πρώην Ε, αν έχουμε για παράδειγμα μια αναθεώρηση μιας υπόθεσης, ποιος θα ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Έχουμε επίσης κάποια θέματα προστασίας μαρτύρων και τα μέτρα πραστησία μπορεί να πρέπει να αρθούν ποιος θα αποφασίσει αν θα έρθουν αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι δικαστική απόφαση και δεν είναι προφανές ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να περάσουν σε διοικητικούς φορείς. Θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση από κάποιο δικαστικό φορέα. Το πρόβλημα αυτό το εξετάζουμε επί του παρόντος. Το εξετάζει και μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και παρά το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση, η ιδέα είναι να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, ο οποίος θα μπορέσει να ασχοληθεί με αυτές τις δομές. Μπορεί να υπάρχουν για παράδειγμα ένας κατάλογος δικαστών και να ε, προσκαλούνται από αυτόν τον κατάλογο αν θεωρείται απαραίτητο. Θα είναι δηλαδή ένας πάρα πολύ ευέλικτος μηχανισμός και οι εκκρεμότητες αυτές θα μπορούσαν ίσως να διευθετηθούν μέσω ενός τέτοιου φορέα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δικαστήριο αλλά και για τη δικαιοσύνη εν γέννη οι δραστηριότητε ενό δικαστηρίου όταν ε, περατώνεται η εντολή του να μην μένουν κενό γράμμα, να υπάρχει μια συνέχεια στην ε, περιοχή. Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό να μιλάμε για στρατηγική ολοκλήρωση και στρατογική συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι η ολοκλήρωση σε διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να έχει μια συνέχεια σε εθνικό επίπεδο και αν θέλουμε το εγχώριο δικαστικό σύστημα να αναλάβει το πρόβλημα και να είναι πραγματικά σε θέση να συζητήσει τα θέματα αυτά και να κάνει δίκες με δίκαιο τρόπο, ε, πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία ήθελα να σας μεταφέρω. Αυτή είναι η δική μας οπτική γωνία και φυσικά είναι ευπρόσδεκτα τυχόν σχόλια για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Ποτσά. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρίτεμπρουκ, η οποία είναι η συγγήτριά μας για τα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστά, κυρίες και κύριοι. Πρωτίστως, νομίζω ότι θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό της Επιτροπής μας, τη γραμματεία της Επιτροπής μας και ιδίως την κυρία Όπατσίτση, η οποία με βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να συντάξω την έκθεσή μου. Δεύτερον θα ήθελα να αναφέρω ότι μαζί με τα τωρινά μέλη του Διεθνούς <clears throat> Δικαστηρίου καθώς και με πρώην μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου έχω συναντήσει μια μεγάλη διαθεσιμότητα να συνεργαστούν μαζί μου, να μεταλαμματεύσουν τις εμπειρίες τους, να εξηγήσουν τι έχουν πράξει. Όλα αυτά είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά και ήταν μια ιδιαίτερα πλούσια εμπειρία το να μπορέσω να εργαστώ με τους δικαστές του δικαστηρίου. Χωρίς αυτούς προφανώς το έργο μου δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί. Θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο δικαστής Πότσερ. Πρώτα απ' όλα όμως να σας υπενθυμίσω τους αριθμούς που εμπλέκονται. Μιλάμε για 161 απαγγελίες κατηγορίας, διαδικασίες που έχουν περατωθεί εναντίον 116 κατηγορουμένων, πολλές άλλες διαδικασίες είναι εν εξελίξη, μόνο 5 κατηγορούμενοι μένουν στο προδικαστικό στάδιο και ξέρετε ότι από όλα τα άτομα στους οποίους κατηγορία, δύο, ο Μλάντιτς και ο εξακολουθούν να μην έχουν συλληφθεί. Το ίδιο το δικαστήριο, όπως ανέφερε ο δικαστής Πόκαρ, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία του να συντάξει ένα σχέδιο το οποίο έχει γίνει γνωστό ως η στρατηγική συμπλήρωσης, υπεράτωσης. Από την αρχή δεν ήταν ποτέ η αρχική πρόθεση το Διεθνές Δικαστήριο να αποτελέσει ένα μόνιμο θεσμό, απλώς να είναι ένας προσωρινός θεσμός στο Δικαστήριο την πρώην με ειδική εντολή και από τη στιγμή που η εντολή αυτή εκπληρούται, το δικαστήριο θα πάψει να υπάρχει. Η βασική λοιπόν ιδέα που διέτρεχε όλες αυτές τις ε, ενέργειες ήταν να γίνει η διαδικασία τις λειτουργίε του δικαστηρίου σε τρία στάδια και ο τωρινός στόχος είναι να συμπληρωθούν όλες οι διαδικασίες, δίκες και ε, ή εφέσεις μέχρι το 2011, το πολύ μέχρι το 2012 και για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα οι τρεις, τα τρία τμήματα τα οποία δικάζουν και το εφετείο εργάζονται επί συνεχούς βάσης. Ναι, τα πρωτοβάθμια τμήματα και το εφετείο. Επίση, οι δύο μη συλληφθέντε για τους οποίους έχει απαγγελθεί κατηγορία αναμένουμε ότι θα συλληφθούν και θα έρθουν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Γιατί δεν πρέπει με το τέλο της εντολής του δικαστηρίου να τύχουν ατιμορρησία. Αυτό αποκλείεται. Είναι πολύ σημαντικό επιπλέον όταν φτάσουμε στο φυσιολογικό πέρας της ε, θητείας του δικαστηρίου να συνεχίσουν οι δίκες να διεξάγονται με την απόλυτη αυτή προσοχή και ενδελέχεια η οποία της έχει χαρακτηρίσει μέχρι τώρα. Δεν πρέπει λοιπόν να διαταραχθεί η πρέπουσα νομική διαδικασία λόγω βιασύνης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το δικαστήριο να εξακολουθήσει να έχει υψηλού επίπεδου προσωπικό. Γιατί μάθαμε ότι σιγά σιγά καθώς πλησιάζει το τέλος της εντολής του δικαστηρίου πολύ υψηλά προσοντούχοι εργαζόμενοι στο δικαστήριο μπορεί να έχουν τον πειρασμό να πάνε να εργαστούν αλλού. Για όλους αυτούς τους λόγους οι συστάσεις μας ζητούν από το Συμβούλιο να εξετάσει κατά πόσο χωρί λόγος για μία παράταση της εντολής του δικαστηρίου για δύο χρόνια, κατά πόσον επίσης θα είναι επαρκής μια διετής παράταση. Ζητούμε από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για να πείσει τις εμπλεκόμενες χώρες να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη σύλληψη των δύο ατόμων που εξακολουθούν να παραμένουν εν ελευθερία παρά την απαγγελία κατηγορίας και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης σημαίνουν το να υπάρχει και μια πλήρως λειτουργούσα δικαστική εξουσία στο κράτος αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει και όλες τις δίκες που έχουν να κάνουν με παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ακόμα και όταν δεν υπάρχει πλέον το πλέγμα των φορέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Παρά το γεγονός ότι κατανοούμε ότι η εθνική κυριαρχία είναι <clears throat> ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς δικαιακού συστήματος, είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να υποστηρίξει την, ανάπτυξη μιας εσωτερικής, μιας εθνικής ικανότητας των δικαστηρίων, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο του διεθνούς δικαστηρίου, τα, εγχώρια δικαστήρια. Υποστηρίζουμε τη συνέχιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων τα οποία έχουν ευρεία εμβέλεια βάσει του μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη στρατηγική της για τη διατήρηση των ενεργειών του Διεθνούς Δικαστηρίου στα ποινικά θέματα και ζητούμε ακόμα πιο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των ανακριτικών αρχών στα Δυτικά Βαλκάνια στις εμπλεκόμενες χώρες, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Γνωρίζουμε επίσης και καταγράφουμε ότι η ύπαρξη ενός σαφούς μηχανισμού για να αντιμετωπίσει τα υπολείποντα, τις υπολείπουσες λειτουργίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα είναι κάτι κομβική σημασία για να εξετάσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι η κληρονομιά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα είναι αυτή η οποία μπορούμε να περιμένουμε βάσει της εντολής τους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι δομές και οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν που θα επιτρέψουν οι υπολοιπόμενες λειτουργίες του δικαστηρίου να εξασφαλιστούν. Αναφέρουμε τις πιο σημαντικές από αυτές τις λειτουργίες που παραμένουν και προτείνουμε να υπάρξει μια πρόταση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ενδεχόμενη δημιουργία ενός κοινού γραφείου που θα αντιμετωπίσει τις υπολοιπόμενες μάλλον λειτουργίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Ρουάντα και του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε και τέλος υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της συνέχισης του Διεθνούς Δικαστηρίου με το ότι τα αρχεία του θα πρέπει να αποθηκευτούν σε κατάλληλη τοποθεσία και τονίσουμε ότι η συνέχεια της ύπαρξη του διεθνού Δικαστηρίου θα πρέπει να συνδέεται με τη διαδικασία συμφιλίωση στις εμπλεκόμενη χώρες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Δικαστά, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτέ είναι οι βασικέ ιδέε ε, του σχεδίου σύσταση που εγώ είχα την τιμή να υποβάλω στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Μέτς. Η κυρία Κάλενμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Πόκαρ για την παρουσίασή σας. Τρία ερωτήματα έχω. Μας περιγράψατε τις ενέργειες που έχετε κάνει ώστε να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική τερματισμού των διαδικασιών και στη συνέχεια να μπορούν τα τοπικά δικαστήρια να αναλάβουν τη σκητάλη. Κάτι το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει είναι η διαρκεία αυτών των ε, διαδικασιών. Στην περίπτωση του Κοτοβίνα και του Σέσελ, παραδείγματος χάρη, είναι διαδικασίες οι οποίες τρέχουν για χρόνια. Σημαίνει αυτό ότι δεν είχατε αρκετή υποστήριξη, δεν είχατε αρκετό προσωπικό. Αυτό θα ήθελα πολύ να γνωρίσω. Και επίσης θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου ότι άτομα τα οποία είναι γνωστά όπως ο Σεσέλη εξακολουθούν να ασκούν δραστηριότητες στη χώρα του, στη χώρα τους ως αρχηγοί κομμάτων παραδείγματο χάρη. Επίσης, όταν αναφέρονται το θέμα της Βοσνίας και του και των ε, διαδικασιών που συνδέονται με τη Βοσνία, υπάρχει πολλές φορές το ερώτημα ότι, ότι για την περίπτωση παραγωγός χάρη ατόμων από το κοσφοπέδιο δεν υπήρξε η ίδια διοκτική ενεργητικότητα κατά κάποιο τρόπο και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το θέμα αυτό. και επίσης θα ήθελα να αποφασιστεί η περίπτωση του Κοντινάη. Ο κύριος Πριμπέτης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον καθηγητή και τη συνάδελφό μου την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο συστάσεως και θα ήθελα υψηλόφωνα να εκφράσω προβληματισμό για δύο πτυχές της εν λόγω συστάσεως. Κυρίως όσον αφορά το σημείο D λατινικό και το G λατινικό. Για το D θα ήθελα να έχουμε μια επέκταση της θητείας του Κοινοβουλίου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και του Ράντοβαν Καράτζιτς και του Γκόραν Χάτζιτς που ήταν επικεφαλής του Σερβικού Στατού στην, ε, στην Κροατία. Διερωτώ με λοιπόν ποια, πώς ερμηνεύονται κάποια ψηφία και σε αιτία του δικαίου. Δηλαδή του Μαΐου του 1913 του 827 του Συμβούλιο Ασφαλείας το 1993 που δεν καθόριζε προθεσμίες για την εντολή που δίνονταν στο δικαστήριο οπότε ήταν μια δίκη, μια διαδικασία αορίστου διαρκεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο ψήφισμά του 1503 του 2003 καθόρισε μια στρατηγική ολοκληρώσεως των διαδικασιών προσπαθώντας να δώσει προσανατολισμό στα δύο ποινικά δικαστήρια για την πρώην Ιγκοσλαβία και τη Ρουάντα θέλοντας στην ε, πρωτοβάθμια φάση και στις υπόλοιπες φάσεις οι δίκε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010. Αυτή η προθεσμία ήταν απλώς ενδεικτική, ένας προσανατολισμός, μια στρατηγική που θα επέτρεπε την αποτελεσματική ε, ολοκλήρωση των δικασιών και ανακοίνωσε το δικαστήριο ότι λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκκρεμούσες δίκες και κυρίως αυτή του Ράντο Βαν Κάρατζιτς ότι δεν θα τηρηθεί αυτή η προθεσμία και μάλλον 2012, τέλος του 2012 ήταν είναι προθεσμία. Δεν αναφερόταν ημερομηνίες, δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Οπότε αυτό το ψήφισμα το 827 ήταν πολύ ισχυρότερο διότι έδινε μια κατεύθυνση, ένα προστατολισμό 2003 καθόριζε σαν ενδεικτική προθεσμία και όχι καταληκτική. Στο πνεύμα των δύο ψηφισμάτων λοιπόν θα πρέπει να παραμείνουμε σε, αυτή την, ε, σε αυτό το πλαίσιο. Να δοθεί ένα κίνητρο, μια παρένεση για να, γίνει σεβαστό, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και των κατηγορουμένων, αλλά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή να υπάρχει κολλησιεργία μέσω της εφαρμογής των δικαιωμάτων και να καθυστερήσουν οι διαδικασίες. Αυτό είναι βασικό στοιχείο στη σύσταση, στην παράγραφο D λατινικό, υπάρχει ένα πρόβλημα λογικό και νομικό θα έλεγα όσον αφορά την σύλληψη των δύο, του πνεύματος των δύο του 1993 και του 2003. Διότι πιστεύω ότι αυτές οι δύο, ε, αυτοί οι δύο σταθμοί επιτρέπουν την καλύτερη ορατότητα του διαβήματος. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάποια ε, προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τους φυγόδικους, για να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των διώξεων αυτών. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά στεναροί, να έχουμε καλή δομή στο ψηφισμά μας. Θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, να αποδοθούν οι ευθύνε και καταδικαστούν, αλλά εγκαίρως οι κατηγορούμενοι. Δεύτερο, ένα σημείο που είναι αρκετά ευαίσθητο και αφορά το σημείο J, το λατινικό, το πρόβλημα των αρχείων, που είναι αρκετά σημαντικό και ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο, διότι αυτά τα αρχεία διαβιβάζονται από τα κάτι μέλη, άμα υπάρχει αίτημα για συνεργασία, και πολύ συχνά κοινοποιούνται υπό την μορφή εμπιστευτικών αρχείων, στη μεγάλη πλειοψηφία τους. Όσον αφορά τα αρχεία ενός οργάνου, ενός φορέα των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να παραμένουν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών αυτά τα αρχεία. Και αυτή η σύσταση θα πρέπει να διευκρινίζει βασικά ότι σίγουρα μπορεί να υπάρχει περιφερειακή μετακίνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό παρά μόνο από έναν όρο. Ότι η διαδικασία θα γίνει υπό την άδεια, την κυρίαρχη και τον έλεγχο του ΟΗΕ. Χρειάζεται μια σχετική τροποποίηση, μια σχετική τροπολογία. Ούτε ώστε να μην δοθεί κακή ερμηνεία αυτή τη πτυχή τη περιφερειακή μετακινήσεω των αρχείων που είναι πάντα ένα ευαίσθητο θέμα σε τέτοιε περιστάσει. Ευχαριστώ. Και τελευταίος στον πρώτο γύρο η κυρία Ντόρις Πακ. Ευχαριστώ κύριε Ποκά. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το οποίο ελήφθη, ελέγχθη από πολλούς, ότι δεν είναι το δικαστήριο το οποίο θα οδηγήσει κατά ανάγκη σε συμφιλίωση αλλά τα πορίσματα του δικαστηρίου, οι αποφάση του ίσως θα οδηγήσουν στο μέλλον σε μια συμφιλίωση μεταξύ των εμπλεκομένων, χωρίς κάποια καταδίκη ατόμων όπως ο Μλάντης και ο Κάρατζης. Δεν είναι δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή της Βοσνίας. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα περισσότερο. Το ένα ερώτημα το έθεσε η κυρία Κάλεμπαχ. Είναι δυνατόν ότι ο Χάσιτς δεν έχει ακόμα ότι ο Σέσελ συγγνώμη, δεν έχει δικαστεί ακόμα και εξακολουθεί να ηγείται ενό πολιτικού κόμματος και να έχει επιρροή σε μια χώρα η οποία θέλει να είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο λογικό χρονικό πλαίσιο για να κλείσει αυτή η διαδικασία. Όλα αυτά μου δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες. Δεύτερον, θέτω αυτό το ερώτημα. Αν τόσο πολύ βραδύνει η διαδικασία με τον κύριο Σέσελη. Πόσο καιρό θα περιμένουμε για να τελειώσει η διαδικασία με τον κύριο Κάρατζιτς. Εγώ θέτω στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα όταν βλέπω πόσο βραδύ είναι αυτή η διαδικασία και συνεχίζω αυτά που είπε ο Γάλλος ε, συνάδελφος. Δεν βλέπω καμία κανένα λόγο να μιλάμε για το τέλος της διαδικασίας αυτού του δικαστηρίου, όταν δεν έχουν κλείσει αυτές τις διαδικασίες. Να πούμε ότι όλα πρέπει να κλείσουν μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορεί να περατώσει το έργο του το δικαστήριο το ποινικό, μέχρι ότου έχει τελειώσει η διαδικασία εναντίον δύο από τους πιο σημαντικούς κατηγορούμενους. Αν κλείσει πια η διαδικασία του δικαστηρίου, θα πούν ορισμένοι στις χώρες αυτές, ε, εντάξει, μόλις κλείσει η διαδικασία, τότε θα ανεβρεθούν αυτοί οι οποίοι αναζητούνται και δεν έχουν συλληφθεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πότε θα μπορέσει να συλληφθεί ο κύριος Μλάντης. Το ουσιαστικό να πάει να έλθει ενώπιον του δικαστηρίου. Θα πρέπει επομένως να επιζητήσουμε το έργο του δικαστηρίου για τα ποινικά θέματα για τα εγκλήματα στην πρώην Ιουκοσλαβία ότι δεν θα πρέπει να περατωθεί. Προφανώς θα πρέπει να κλείσουν οι διαδικασίες αυτές οι οποίες είναι εξελίξη, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες εναντίον αυτών οι οποίοι ακόμα δεν έχουν δικαστεί. Και έχω ένα ακόμα πράγμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Θα μπορούσατε να μας δώσετε τη δική σας εντύπωση που έχετε αποκομίσει από τα δικαστήρια τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες πολέμου στην ε, περιοχή. Έχω μιλήσει με τους υπευθύνους στο Βελιγράδι και ήταν ήδη πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ εντυπωσιακή η εργασία τους για τα θέματα της δίωξης των εγκλημάτων πολέμου. Μπορείτε να πείτε κάτι αντίστοιχο για τη Βοσνία Ζεχοβίνη. Υπάρχουν ε, ελλείψεις για τα θέματα αυτά δίωξη των εγκληματιών πολέμων. Μπορείτε να δακτυλοδεικτήσετε τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή σε ό,τι αφορά τι δικαστικέ αρχέ για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά. Μιλήσατε επίση και για μνημεία, για χώρου ενθύμηση. Μπορείτε να μα πείτε κάτι περισσότερο για τα Βαλκάνια και του χώρου αυτού ενθύμηση. Κύριε καθηγητά, τέθηκαν πολλά ερωτήματα. Θα μπορούσατε να απαντήσετε σε κάποια τουλάχιστον από αυτά σε αυτό το πρώτο γύρο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις που θέσατε. Και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια που εξήγησε το περιεχόμενο του σχεδίου συστάσεως που ετοιμάζεται για το Συμβούλιο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για εκρεμείς υποθέσεις. Δεν μπορώ ως δικαστής να σχολιάσω εκρεμείς υποθέσεις. Μπορεί να φτάσουν στα χέρια μου και να μην είμαι μέλος. Υπάρχουν πολλές ε, προσφυγές που μπορεί να γίνουν. Εγώ είμαι στον ε, δεύτερο βαθμό. Δεν θέλω λοιπόν να εμπλακώ σε σχολιασμό εκκρεμουσών υποθέσεων είναι αντιδιοντολογικό σε σχέση με την αρμοδιότητά μου ως δικαστού. Πρώτον, η διάρκεια των δικών, εν γέννη. Όταν πήγα κι εγώ στο δικαστήριο, πραγματικά ξεπλάγινα από την διάρκεια κάποιων υποθέσεων. Κατόπιν άρχισα να το καταλαβαίνω κι εγώ. Γιατί κρατούν τόσο οι δίκες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν τα εθνικά δικαστήρια. Διερμηνία, μετάφραση. Ε, η δίκαιη δίκη απαιτεί να μπορεί ο κατηγορούμενος να διαβάσει το υλικό. Στην ακρόαση έχουμε διερμηνείς στην ε, ακροματική διαδικασία. Τα γραπτά κείμενα ωστόσο πρέπει να μεταφραστούν. Ο εισαγγελέα μιλά και γράφει κάποια κείμενα σε μία γλώσσα. Η υπεράσπιση γράφει και μιλά σε άλλη γλώσσα. Η γλώσσα της δίκης είναι αγγλικά ή γαλλικά, πέραν των ε, Σερβοκράτικων βεβαίως, διότι ε, οι μάρτυρες ε, μιλούν κατά βάση τη γλώσσα τους. Και μερικές φορές έχουμε και τα Ολλανδικά. Χρειάζεται λοιπόν μετάφραση. Και καλή μετάφραση των κειμένων. Εξού και εν μέρη η καθυστέρηση. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της συνεργασίας των κρατών. Πρόκειται για την πρώτη φορά δεν συνέβαινε αυτό στην Εμβέργη, που δημιουργείται ένα διεθνές δικαστήριο και χρειάζεται να στηρίζεται στη συνεργασία των χωρών. Δεν έχει δηλαδή τον έλεγχο στην, στον χώρο όπου έγιναν τα γεγονότα που δικάζει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας συνδυασμός των απαιτήσεων ενός δικαστηρίου με τις απαιτήσει που έχει ένα κράτο από την αίτηση ε, δικαστική συνδρομή που ένα κράτο κάνει σε ένα άλλο κράτο, σε μια άλλη υπόθεση. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δικονομικέ καθυστερήσει που υπάρχουν ακόμα και όταν υπάρχει προθυμία συνεργασίας ενός κράτους. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Εξού και μία αιτία καθυστέρησης. Ένας άλλος λόγος που αντιμετωπίζουμε και στα εθνικά δικαστήρια είναι ότι οι εγγυήσει που πρέπει να παράσχει ένα διεθνές δικαστήριο είναι μερικές φορές ε, μεγαλύτερα, μεγαλύτερες από αυτές τις απαιτήσει που απαιτούνται σε ένα εθνικό δικαστήριο. Ξέρετε ότι η έννοια της δίκαιης δίκης σε διεθνές επίπεδο κάθε διεθ... βρίσκονται και περιγράφονται σε κάθε διεθνές κείμενο ως ελάχιστες εγγύησεις. Μερικές φορές τα κράτη-μέλη τηρούν αυτές τις ελάχιστες εγγυήσεις. Ένα διεθνές δικαστήριο πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη εχέγγυα. Επίσης, υπάρχει το θέμα της προστασίας των μαρτύρων που είναι συχνά θύματα. Πρέπει να τους μεταφέρουμε στη Χάγη, να εξασφαλίσουμε ότι όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους δεν θα υποστούν κάποια είδη αντιπίνων. Ένα δύσκολο πάντα ζήτημα. Και μάλιστα πολλοί μάρτυρες δεν ξαναγυρίζουν πίσω πηγαίνουν αλλού με άλλο όνομα και εξαφανίζονται, δηλαδή ξεκινούν μια νέα ζωή κάπου αλλού γιατί είναι πολύ δύσκολο για τα άτομα αυτά να γυρίσουν πίσω. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι παράγοντες που τα εθνικά δικαστήρια δεν αντιμετωπίζουν και καθιστούν ε, μεγαλύτερες, μακρύτερες τις διαδικασίες αυτές. Βεβαίως προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τις δικαστικές διαδικασίες υπό τον όρο της στήριξης της αρχής της δίκαιας δίκης. Δεν θέλουμε να αφησιάσουμε οποιαδήποτε αρχή δίκαιης δίκης για να τηρήσουμε την στρατηγική περάτωσης, για παράδειγμα. Αυτό το έλεγα πάντα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. υπάρχει και ένα ζήτημα της αμεροληψίας που δεν θα φύγει. Εγώ πιστεύω ότι το δικαστήριο είναι αμερόληπτο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση, η κάθε μάλλον απόφαση, λαμβάνεται από τους δικαστές βάσει των μαρτυριών και αν και μόνο. Αν έρθουν τα αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο θα τα λάβουμε υπόψη. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία για τον ΑΒ λόγο δεν φτάσουν στα χέρια μας, η μόνη επιλογή που έχουν οι δικαστές είναι να στηριχθούν στα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν. Τώρα, η βάση, ο λόγος της περάτωσης, όντως το βασικό κείμενο του ΙΕ δεν έθετε η ημερομηνία. Πρωτοβουλία του δικαστηρίου ήταν να ξεκινήσει όχι μια ημερομηνία αλλά μια στρατηγική πιθανής ημερομηνίας. Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000 δεν είχαν δείξει οι ασκήσεις δίωξης. Το 2004 έλεξαν και είχαμε αναρωτηθεί πόσο χρόνο θα θέλαμε για να αντιμετωπίσουμε όλα όσα ήθελε ο εισαγγελέα να κρίνει. Και είχαμε πει ότι με τα στοιχεία θα κλείναμε το 2016 και αποφασίσαμε ότι το 2016 παρά ήταν μεγάλο, μεγάλος χρόνος γιατί χάνονται οι μάρτυρες, πεθαίνουν. Οι κατηγορούμενοι επίσης πεθαίνουν. Είναι δύσκολο να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία τόσο πολύ πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα και αποφασίσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Για να παρουσιάσουμε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας είπαμε ο χρόνος που απαιτείται είναι υπερβολικά πολύ, πρέπει να τον περικόψουμε ενδεχόμενα και κατά 50%. Γι' αυτό ε, έφτασε η ημερομηνία του 2008, αλλά ζητήσαμε να αυξηθεί, να διπλασιαστεί ο ρυθμός των δικαστών. Έτσι βγήκε το, η, χρονολογία. Ήταν μια ε, ασαφής εκτίμηση καθυπολογισμών όταν είδαμε πόσες ε, διώξεις θα ασκούνται Τώρα, όταν σταμάτησαν ε, να, να κατηγορίες το 2004, ε, είχαμε τους 261 και λάβαμε υπόψη και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και είδαμε ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε αν συλληφθούν οι δύο φυγόδικοι. Σύντομα να κλείσουμε, λέγαμε γύρω στο 2011-12. Αλλά και πάλι πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της δίκης δίκης. Δεν μπορούμε να επιταχύνουμε πολύ την κατάσταση και οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε βελτιώσανε τους δικονομικούς κανόνες προσκόμιση στοιχείων και μαρτυριών αλλά και πάλι χωρίς να φύγεται η δίκαιη Το, για το θέμα της ε, συμφιλίωσης είπα ότι το ε, δικαστήριο μόνο να βοηθήσει μπορεί την ε, συμφιλίωση στην περιοχή. Δεν μπορεί μόνο του να παρέμβει. Αλλά για να υπάρξει εμφυλίωση πιστεύουμε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη από το δικαστήριο πρέπει να δικαστούν από το δικαστήριο. Κάποιες περιπτώσεις δεν τις εξετάσαμε γιατί ήταν μικρά αδικήματα, αλλά ε, υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις που ήδη τα ίδια τα εθνικά δικαστήρια θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να τα κρίνουν ε, σωστά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το δικαστήριο πρέπει να είναι εκεί όπου έγιναν τα γεγονότα, γιατί η απόφαση εκεί έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και στον πληθυσμό και εξυπηρετεί περισσότερο και τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Πρέπει ωστόσο να γίνονται, σεβαστά κάποιες, να γίνονται σεβαστές κάποιες εγγύησεις. Πιστεύω ότι τα δικαστήρια εκεί δουλεύουν σωστά. Έχουμε την εμπειρία μεκτών δικαστηρίων στο Σεράγεβο που ήταν μια καλή εμπειρία. Έγιναν δικαστήρια, ε, πολλά, πολλές ε, δίκες έγιναν με μεικτά δικαστήρια και με τη βοήθεια ε, δικαστών εξωγενών από το μερικών από τους οποίους και από το δικό μας δικαστήριο. Τώρα για αυτά τα κέντρα μνήμης Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται να, υπάρξει, να υπάρξουν τέτοια κέντρα και για σκοπούς συμφιλίωσης και μόνο, για να βοηθήσει γενικά τον πληθυσμό να καταλάβει τι έκανε το δικαστήριο και γιατί αποφασίστηκε αυτό ή εκείνο στην ΑΒ δίκη. Είναι σημαντικό για κάποιον που δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι ειδικό σε τέτοια θέματα, να μπορεί να καταλάβει σωστά την απόφαση του δικαστήριο. Προφανώ χρειάζεται κάποια βοήθεια. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε στο κομπιούτερ και να του πούμε διάβασε το υλικό και θα καταλάβει. Πρέπει να έχει κάποιου πιο ειδικού που να εξηγούν στον κόσμο πώ να διαβάσουν τα κείμενα και να καταλάβουν. Και να καταλάβουν επίσης ότι κάποιες αποφάσεις οφείλονται στα στοιχεία που είχε μπροστά του στα χέρια του δικαστήριου. Το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν και που δεν είναι κατά ανάγκη Ταυτόσιμα με τα γεγονότα, αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Δεν είναι 100% αυτό που έγινε, αλλά αυτά που έφτασαν στα χέρια του δικαστήριου. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ τρεις, τρεις ακόμα μιλητές. Η κυρία Γκόμης. Κύριε Πόκαρ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Ανεμή για τη θαυμάσια εργασία που έχει κάνει και συμφωνώ και με πολλές από τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεσή της ίσως όχι όλες. Θα ήθελα τώρα να προτείνω να λάβει υπόψη η κυρία Νέιτς την δυνατότητα να ενημερώσει την εκθεσή της κάνοντας και μία μνήα των ε, προσφάτων δηλώσεων που έκανε ο αρχισαγγελέας Μπράματς όταν επισκέφθηκε την Κροατία την προηγούμενη εβδομάδα και τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά τεκμήρια για την δίκη του Άντρα Ιγκοτοβίνα που δεν έχουν ακόμα παραδοθεί από την κυβέρνηση της Κροατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επειδή θα υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Κροατίας αύριο, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο φυσικά μπορούμε να εγείρουμε αύριο και εγώ θα το πράξω, αλλά σίγουρα αυτό θα πρέπει να ληφθεί στην έκθεση υπόψη. Τα ερωτήματά μου τώρα <clears throat> είναι τα εξή. Πώς εσείς ως δικαστής κύριε Ποκάρ θεωρείτε μπορούμε να διατηρήσουμε ε, τον ρυθμό που έχει επιτύχει το δικαστήριο για τη σύλληψη και των υπολείπων κατηγορουμένων. Αν βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση περάτωσης ή ολοκλήρωση των εργασιών του δικαστηρίου, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Θα πρέπει να μην δικαστούν αν έχει κλείσει ουσιαστικά το δικαστήριο μήπως θα πρέπει να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από το Συμβούλιο Ασφαλείας και επίσης οι λεγόμενες υπολοιπόμενες λειτουργίες του δικαστηρίου πέραν των προτάσεων της ανεμίας. Όχι μονάχα για αυτό το δικαστήριο αλλά και για τα άλλα προσωρινά δικαστήρια της Σιέρα και τη Ρουάντα. Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα μιας ε, λύσης βάσει της οποίας θα υπάρξει παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ώστε να αναλάβει τα υπολοιπόμενα εγχειρήματα επί τη βάση ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας βέβαια. Ο κ. Μπίστλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλά από αυτά που θέλω να πω έχουν καλυφθεί και ζητώ συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι. Αλλά μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκόμες, εγώ θέλω να στραφώ προς, τον, προς την εισηγήτρια και όχι προς τον καθηγητή Πότσαρ. Στην έκθεσή της αναφέρει τα, την περίπτωση δύο κατηγορουμένων οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ερημοδικία, για να δικαστούν ερήμην αυτοί οι δύο και να καταδικαστούν εάν θεωρηθούν ε, ένοχοι. Αλλιώς μήπως θεωρεί η συγγήτρια ότι θα ήταν σκόπιμο να προτείνει πράγματι να λάβει χώρα η δίκη για τα δύο αυτά άτομα. Και τέλος η κυρία Όμεν Ρέιτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νέιτς για την έκθεσή της είναι ιδιαίτερα λογική. Είναι σαφές ότι το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο με 116 υποθέσεις έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και μπορεί να παρουσιάσει και πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν ε, σημαίνει κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό μάλλον το γεγονός ότι παραμένουν και κάποιοι ε, ελεύθεροι και δεν έχουν ακόμα δικαστεί, αλλά Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέει η κυρία Νέιτς για την πλήρη συνεργασία με το ποινικό δικαστήριο από τις χώρες στις οποίες υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία διαφεύγουν της δίκης και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δεσμευτεί σε αυτή τη συνεργασία. Δεν θα ήμασταν λοιπόν αξιόπιστοι εάν δεν τηρούσαμε τις δεσμεύσεις μας. Η αξία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι τόσο μεγάλη ακριβώς γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανακοδόμηση του δικοστικού συστήματος ε, στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα από τα βασικά κριτήρια της ε, Κοπενχάγης, επομένως την χάνει της ε, μέγιστης προσοχής μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα λέει η κυρία Νέιτ στην έκθεσή της και ε, για το σημείο του κληροδοτήματος που θα αφήσουμε στα δικαστήρια ε, το θέμα της, ε, συνεχής, της συνεχούς πορείας της Έχω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Οι προθεσμίες. Προφανώς την απόφαση τη λαμβάνουν τα, τα Ηνωμένα Έθνη. Προφανώς και το δικαστήριο θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί μετά το 2010. Αλλά αυτή τη στιγμή καθορίζεται μια καταληκτική προθεσμία. Σημαίνει ότι οδεύουμε προς το τέλος. Εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε μια πιο αμφίσιμη, να μην έχουμε τόσο αμφίσιμη ε, ερμηνεία και να μείνουν ε, ε εκρεμείς υποθέσεις. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευ... ευέλικτα τα πράγματα προς την ημερομηνία. Η κυρία Νέιτς λέει πολύ σωστά ότι ε, όταν ε, ε, βγαίνει η απόφαση ενός δικαστηρίου δεν σημαίνει ότι τελειώνει και το καθήκον του δικαστηρίου. Κάποια στοιχεία που έχουμε μάθει, οι καλές και κακές μας εμπειρίες από το δικαστήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εμπειρία θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω ε, από την εισηγήτρια πώς σκοπεύει να εισαγάγει αυτά τα στοιχεία στο κείμενό της. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον καθηγητή Ποσάρο, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις σας και μετά ε, η κυρία Νέιτς θα ολοκληρώσει. Παρακαλώ, καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Δεν θα απαντήσω φυσικά στις ερωτήσεις που στρέφονται προς την εισηγήτρια. Για το Βλάντιτς και το Χάτζιτς. Τι θα γίνει αν το δικαστήριο κλείσει πριν τη σύλληψή τους. Η θέση που υποστηρίζει πάντα το δικαστήριο είναι ότι οι δύο αυτοί οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν στη Χάγη. Ή θα πρέπει να δικαστούν από τον ε, μηχανισμό αντιμετώπισης αυτών των εκκρεμών υποθέσεων που θα μείνει. Θα πρέπει λοιπόν πίσω από αυτό το μηχανισμό θα πρέπει να, ε, να υπάρχει και η δυνατότητα για έναρξη μιας νέας δίκη για κατηγορημένους οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί πριν από τη λήξη της θητείας του δικαστηρίου. Εάν ε, συλληφθούν πριν από το κλείσιμο του δικαστηρίου θα υπάρξει υποθέτω κάποια παράταση για την στις ε, δύο αυτές υποθέσεις. Όχι για όλα τις υποθέσεις, αλλά για να μπορέσουν να περατωθούν αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, το να παραπευθούν αυτές οι υποθέσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι πρόκληση, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο υπάρχει και έχει αρμοδιότητες οι οποίες δεν ε, αφορούν μια στενή γεωγραφική έννοια. Το πρόβλημα όμως είναι νομικό. Υπάρχει ένα νομικό κόλλημα. Το ίδιο το καθεστώς του δικαστηρίου μιλάει για δικαιοδοσία του δικαστηρίου μόνο για εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν μετά από την 1η Ιουλίου του 2002. Από τότε ισχύει ο ιστορικός κανονισμός. Και τα εγκλήματα αυτά έχουν διαπραχθεί προ αυτής της ημερομηνίας. Όταν μια υπόθεση παραπέμπεται στο Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο από το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, υπάρχει ένα νομικό άνοιγμα και λέει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωμένη ε, να τηρήσουν τον κανονισμό. Αλλά υπάρχει και η άλλη φιλοσοφική σχολή, αν θέλετε, που λέει ότι το δικαστήριο θα πρέπει να σεβαστεί τον κανονισμό του. Η μόνη περίπτωση στην οποία υπήρχε ε, παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το Συμβούλιο Ασφαλείας πρόσεξε ιδιαίτερα και στην απόφαση παραπομπής έλεγε ότι ισχύει μόνο για εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν μετά από την 1η Ιουλίου του 2002. Σαφώς λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ήθελε να φέρει αυτό το πρόβλημα ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αφήνω όμως το ερώτημα αυτό ανοιχτό. Ως προς το κατά πόσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα ήταν ένας φορέας που θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις εκκρεμότητε, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Αντί να συστήσουμε ένα νέο μηχανισμό, θα μπορούσε το Διεθνές ε, ε, Ποινικό Δικαστήριο να λειτουργήσει ως ένας ε, διοικητικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες όχι μόνο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Κοσλαβία αλλά και για τη Ρουάντα και για τα υπόλοιπα και με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες στις διάφορες περιπτώσεις πότε πρέπει να έχουμε... Ε, ένα μητρό για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ιουγκοσλαβία ή για τη Ρουάντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν βέβαια τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή θα μπορούσε να προσθεθεί ένα επιπλέον πρωτόκολλο στην υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ε, από τεχνικής πλευράς βέβαια είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ως δυνατότητα. Ε, όσον αφορά τις δίκες ερήμην. Το δικαστήριο ήταν πάντα της άποψης ότι δεν θέλει να δικάσει άτομα ερήμην. Τεχνικώς βέβαια υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά εγώ δεν ξέρω κατά πόσον η δίκη ερήμην θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς ε, της δικαιοσύνης περισσότερο από μία παραπομπή. Διότι υπάρχουν ε, κατηγορούμενοι που έχουν παραπευθεί, δεν έχουν ε, συλληφθεί. Σαφώς θα πρέπει να κρύβονται για να μην συλληφθούν. Η καταδίκη ερήμην θα τους δώσει κάτι παραπάνω. Η δίκη ούτως ή άλλως θα πάσχει από κάποιες πλευρές δεν ε, χρησιμοποιήθηκε ποτέ η δυνατότητα από το, αυτή από το δικαστήριο, παρόλο το γεγονός ότι υπήρχε, ε, συνήθως προτιμούμε να έχουμε ενώπιόν μας τον ε, υπόδικο. δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι δύο φυγόδικοι κατά την άποψή μας θα πρέπει να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία ή το μηχανισμό ο οποίος θα συσταθεί κατόπιν της λήξης της αιτίας του δικαστηρίου. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, να αποσταλεί μήνυμα από τα Ηνωμένα Έθνη ότι μένουν ατιμόρυτοι και ότι δεν έχουν δικαστεί έγκαιρα. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. you, Ευχαριστώ καθηγητά. Κυρία Μέιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην διεξαγωγή της συζήτησης και τον δικαστή Πόκα που εμπλούτησε τη συζήτηση με την εμπειρία του και τη σοφία του και τις γνώσεις του. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τι ευχαριστίε μου επισημένοντα ότι και εγώ ωφελήθηκα από την ε, συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών και τη βοήθεια του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοιμάζοντας την έκθεση. Να πω στους συναδέλφους ότι θα εξετάσω τι πιθανότητες υπάρχουν, να λάβω υπόψη τις τάσεις, θα υποβάλω δύο τροπολογίες που αφορούν το δικό μου σχέδιο ψηφίσματος, μια πράγματι θα αφορά την έλλειψη συνεργασίας από την Κροατία, διότι αυτό είναι κάτι καινούριο, το ακούσαμε προημερών. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Και δεύτερον, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι δύο ε, κατηγορούμενοι των οποίων απαγγέλθησαν κατηγορίες θα πρέπει να δικαστούν είτε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην ή από τον επικουρικό μηχανισμό που προβλέπεται. Τώρα για την ερημοδικία ε, δόθηκε απάντηση όσον αφορά του πόσο, κατά πόσο θα ήταν ευκταίο. Θα απαντούσα παρομοίως αλλά είναι πλέον αρμόδιος ο κύριος δικαστής και απάντησε. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους. Να τους επενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 17 Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε πρώτα στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Κοινοβουλίου του Μαρτίου. Ακριβώς. Έχετε μία εβδομάδα, λέει ο Πρόεδρος, για να υποβάλλετε τις τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον δικαστή Ποσάρ και την εισηγητριά μας και όλους σας. Και τώρα θα πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα ενάπτυξη σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Άντριου Ντάφο συντάκτης του κειμένου είναι εδώ και δίνω το λόγο στον ε, Άντριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σε όλους. Όπως ε, ξέρετε μου ζητήθηκε να συντάξω μία γνωμοδότηση για την έκθεση της ε, ΑΦΚΟ, της Επιτροπής. Ο αξιότιμος συνάδελφος ο κ. Μπροκ τα ανέθεσε και θέμα ήταν η αυξανόμενη σημασία των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις ε, προοπτικές ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κ. Μπροκ σήμερα το απόγευμα είναι ενώπιον του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Καλσρούη, προασπιζόμενος τη συνθήκη σε μια υπόθεση που εκδικάζεται στο δικαστήριο αυτό και ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Είναι σημαντικό, πιστεύω, ευθύς εξ αρχής να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται περί διαγωνισμού μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πρόκειται περί ανταγωνισμού για τον έλεγχο της κοινή εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Και είναι σημαντικό εμείς εδώ που είμαστε συγκριτικά νέοι στον τομέα αυτό της ΚΕΠΑ να εκτιμήσουμε τις ευθύνες που υπέχουν τα εθνικά κοινοβούλια. σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Θα πρέπει επίσης όμως να πούμε με κάθε εμπιστοσύνη και πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο έχει αυξανόμενη σημασία όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφαλείας και τα συναφή προβλήματα και προκλήσεις και τη διαμόρφωση σχετικής πολιτικής. Και ο ρόλος που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά κεντρικός. Έχει μεγάλη σημασία για την ε, αύξηση της εμπιστοσύνης στην ΚΕΠΑ. Και ότι αυτή διαμορφώνεται με δημοκρατικό τρόπο. Πρέπει να συμπεράνουμε λοιπόν ότι είναι ε, επικουρική η λειτουργία μας και θα πρέπει να συνεργαστούμε παράλληλα για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε δύο ιδιαίτερες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα μας απασχολεί η χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας από μας φέρει άμεση ευθύνη. όσον αφορά τις δαπάνες για τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών. Και κάτι, το δεύτερο που μας απασχολεί ιδιαίτερος, είναι ότι χρειαζόμαστε όλοι τη σωστή, να φροντίσουμε για τη σωστή ενημέρωση του κοινού. Να υπάρξει εκτίμηση από πλευράς της κοινή γνώμης των προσπάθειών που καταβάλλονται. που πολλές φορές η κοινή γνώμη δεν είναι ενημερωμένη σωστά και δεν εκτιμά σωστά την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην εξωτερική πολιτική. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν σημαντικές ευθύνες. Πρέπει να δράσουν ως δίωδος, ως αγωγός, διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ημών, με ήτα και των εθνικών δημοσίων υπηρεσιών, εθνικών πολιτικών κομμάτων και του τύπου στα κράτη-μέλη. Γιατί για την ώρα δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τη στιγμή που θα υπάρχει αναβαθμισμένη η θέση του Υπουργού Εξωτερικών και ο κύριος Σολάνα θα διοριστεί αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δημιουργηθεί υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα χρειαστεί και καλύτερος έλεγχος της ΚΕΠΑ. Εμείς θα ελέγχουμε την υλοποίηση της πολιτικής αυτής. Θα αυξηθεί ο ρόλος μας. Εκθετικά μάλιστα. Και θα πρέπει ο αναβαθμισμένος Σολάνα, αυτή η φιγούρα, η αναβαθμισμένη του Σολάνα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτροπος. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. αλλά αυξάνεται και η εξουσία ελέγχου που θα διαθέτουμε. σχετικά με τα όσα θα κάνει. Θα πρέπει να προσέξουμε και κάποιες παραγράφους της νομοδοτήσεως. Μάλλον σε κάποιες παραγράφους τονίζω το ότι πρέπει να προσέξουμε τη δική μας θέση εντός των πολυμερών βημάτων συζητήσεων που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των δεκαετιών. Επαναλαμβάνω. Αυτά που είπε το Κοινοβούλιο σε γνωμοδότησή του. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε θέση ισχύ για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, άμα λήξει η θητεία αυτής, θα πρέπει η εμπειρία να διαδοθεί και στα 27 κράτη-μέλη της Δικοπροδικής Ένωσης. Και η διακοινοβουλευτική διάσταση της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση μας εντός της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του ΝΑΤΟ. Είναι ένα χαρακτηριστικό της εκθέσεως Βάτανεν. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, κατά την άποψή μου. Και το επαναλαμβάνω και εδώ. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του πολλαπλασιασμού των άλλων πολυμερών φορέων που αναπτύχθηκαν. Ανέφερα, αναφέρω τρεις τέτοιους φορείς στην παράγραφο 10, αλλά συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί και άλλος φορέας τώρα. Στην Ανατολή. Με τους εταίρους μας της Ανατολικής της πολιτικής μας γειτονίας με τις ανατολικές χώρες. Και πιστεύω ότι κάποιος από αυτούς τους φορείς, από αυτά τα βήματα συζητήσεων, είναι πιο λειτουργικά από κάποια άλλα. Όλα τα βήματα αυτά συζητήσεων μας αυξάνουν το βάρος που επομιζόμαστε. σαν μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά είναι και προς το βάρος και για το προσωπικό μας και για τον προϋπολογισμό μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εξετάσουμε με κριτικό μάτι να κρίνουμε κατά πόσο αξίζουν λοιπόν αυτοί οι φόρεις. και να συγκρίνουμε τους φορείς αυτούς με την μεικτή παραγματος χάρη, με τις μεικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές κλπ. Με άλλους φορείς που έχουμε δημιουργήσει. Κλείνω προτείνοντας το εξή Να επισημοποιήσουμε τις διαιτήσεις αυτές τις διασκέψεις που γίνονται μεταξύ της Επιτροπής μας, που γίνονται δύο φορές το χρόνο μάλλον, και με εκπροσώπους των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν αναφέρομαι μόνο στους προέδρους αυτών των Επιτροπών, αλλά στους συντονιστές που θα έρχονται από τα 27 κοινοβούλια και πολύ συχνά και από άνω και κάτω βουλή. Είναι επιτυχής αυτή η προσέγγιση. Θα μπορεί η επιτυχία να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν η προσέγγιση γίνει συστηματικότερη και αν εντός του Κοινοβουλίου μπορούμε να συλλέξουμε και να αυξήσουμε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, κυρίως σε θέματα ασφαλείας και άμυνας. Έτσι, θα είμαστε αξιοσέβαστοι συνομιλητές για τους ομολόγους μας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι ο κύριος Μπροκ και εγώ θα συμμετάσχουμε στην Κόζακ, στην Πράγα, πριν διακόψουμε τις εργασίες μας για τις εκλογές, για την προεκλογική εκστρατεία και αν περάσει το κείμενο από την Επιτροπή ΑΦΕΤ θα είναι καλό και ενδεδειγμένο να εκφράσουμε τις απόψεις αυτής της Επιτροπής στην ΚΟΣΑΚ. Αυτά έχω να πω. Κύριε Πρόεδρε. Now, uh, I ask Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βλέπω όσου θέλουν το λόγο. Κύριε Ομενρόιτεν. Ορίστικος όδης. και νομίζω ότι πρέπει να διαπραγματευτώ με τον κύριο Νταφ και είναι καλό αυτό γιατί συνήθως συμφωνούμε πάντα. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Καταρχάς, πρόεδρε, το γεγονός ότι δίνει γνωμοδότηση η Επιτροπή Εξωτερικών υπερθέσεων είναι ένα καλό μήνυμα. Ήδη εξορισμού. Από τη στιγμή που η συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ, πρέπει να έχουμε στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί θα έχουμε ε, και άλλες ευθύνες. Θα έχουμε ευθύνη για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα υπάρχουν και εθνικοί βουλευτές, οι οποίοι θα θέλουν και δικαίως να πούν κάτι, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και των εθνικών βουλευτών. Έχουμε λοιπόν κοινέ ευθύνε, οφείλουμε να λειτουργήσουμε ως ο μακρύς βραχίωνας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Έτσι πρέπει να τα δούμε τα πράγματα πρόεδρε. Και αυτό προκύπτει άλλωστε και από το κείμενο του κύριου Νταφ. Επιπλέον, αυτό που δεν είμαι σίγουρη είναι ότι τονίζει πολύ τη συνεργασία στα πλαίσια της Κόζακ. Ε, η Κόζακ αυτή καθ' αυτή είναι λίγο μυστήριο θέμα, όλοι ξέρουμε τι είναι, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Ε, Ούτε εμεί ξέρουμε τι κάνουμε από πλευρά μα ούτε οι εθνικοί βουλευτέ ξέρουν τι γίνεται στην Κόζακ ακριβώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ε, συμφωνίες για τον τρόπο λειτουργία τη Κόζακ. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση. Μιλάμε για συνεργασία, για την ανάγκη να είμαστε ο βραχίωνας ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο οικονομικού ελέγχου. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Όχι μόνο ε, μία συνάντηση το χρόνο με τους ε, εθνικούς βουλευτές, τους φέρνουμε εδώ και κουβεντιάζουμε. Πρέπει να υπάρξει μία μικρή δομή Είχαμε κάτι τέτοιο στους παλιότερες διαβουλεύσεις με τους εθνικούς βουλευτές. Χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει μια ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Τούτο θα είναι θετικό για την εξωτερική πολιτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε σημαντικότερη ευθύνη στον τομέα αυτό. Αυτά ε, θα μιλήσω με τον εισηγητή και δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει η κυρία Ιμπάσκοβα, μάλλον θα συμφωνήσει μαζί μου. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ξέρετε ότι είμαι, βλέπετε ότι είμαι μάλλον ο μόνος σοσιαλιστής εδώ. Ξέρετε, συγγνώμη, ο κύριος Τζολάινεν ζήτησε από τον κύριο Σεβερίν που έφυγε και που μου ζήτησε εμένα να παρουσιάσω τις απόψεις του ως σκιώδους εισηγητού. Ε, συγγνώμη γι' αυτό. Θα σας πω αυτά που λέει ο κύριος Λάιενεν. Υποστηρίζει βεβαίως τα λογικά συμπεράσματα της κατάστασης, δηλαδή ενίσχυση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί αυτοί, αυτά έχουν την ευθύνη του ελέγχου στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα ωστόσο, ε, χρησιμοποίηση των ευκαιριών που έχουμε όσο περισσότερο γίνεται μέσω του προπολογισμού και δεν ξέρω αν το ξέρετε όταν τεθεί ισχύ η Λισαβόνα ε, τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον, αντιπρόσωπο πρόεδρο της Επιτροπής ε, των Μελλοντικών Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης. Ταυτόχρονα ο κύριος Λάινεν πιστεύει ότι θα πρέπει να βγάλουμε μία λέξη από την, τρίτη, από την τρίτη παράγραφο που αναφέρει ότι πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μείζωνα ρόλο στην επίδραση και τον έλεγχο της επερχόμενης ΚΕΠΑ και ΕΠΑ, αρμοδιότητα που μπορεί να συνισχυθεί μόνο με την στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια. Πιστεύεις ότι το only, μόνο, πρέπει να φύγει. Λέμε λοιπόν να ενισχυθεί με την ε, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτές είναι οι, παρα... οι παρατηρήσεις του. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Ιμπάσκοβα. Αυτή τη φορά δεν μπορείτε να ξεφύγετε, θα τα πείτε. Μα δεν είναι πρόκειτο να ξεφύγω. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, με γνωρίζετε εδώ και πέντε χρόνια ότι δεν εκπροσωπώ τα συμφέροντα της δικής μου χώρας και ούτε θα το πράξω τώρα. Αλλά, παρόλα αυτά, η χώρα μου αυτή τη στιγμή προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο εβδομάδες πριν από την έλεξη της Προεδρίας, ο Πρωθυπουργός μου ανέφερε ότι θα κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας από το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Όταν ήρθε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Πρωθυπουργό μου στις 16 Ιανουαρίου, αν δεν απατώμε, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει η κύρωση στο Τσεχικό Κοινοβούλιο μέσα σε δύο εβδομάδες. Πέρασαν τρεις εβδομάδες μετά από αυτή την ομιλία και τώρα λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αιχίας, χρειαζόμαστε ένα και δύο και τρεις μήνες για να το πετύχουμε αυτό. Γίνεται τώρα η συνεδρία της ΚΟΣΑΚ στο, στην Πράγα, ξέρω ότι είναι εξόχως πολιτικά ευαίσθητο το θέμα αυτό, αλλά θα είναι πραγματικά θετικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση σε ένα θετικό και επικοδομητικό πνεύμα για να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Τσεχικού Κοινοβουλίου για να υπάρξει μια ομαλή κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να ενισχυθούν οι εξουσίες και του Τσεχικού Κοινοβουλίου στην, ε, ε, στην ΚΕΠΑ και την ΕΜΑΕ για να μπορούμε να έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποστολές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας όλα αυτά γιατί είχαμε μια αρκετά διαρθρωμένη συζήτηση στο Τσεχικό Κοινοβούλιο τις πρόσφατες εβδομάδες για το Κωσυχοπαίδιο και το Αφγανιστάν και επίσης υπήρξαν και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την συνθήκη της Λισαβόνας που <clears throat> δεν ήταν στον σωστό χώρο διότι είπαν ότι δεν είχαν λόγω της μη κύρωσης συνθήκης της Λισαβόνας τη δυνατότητα να στείλουν πιο πολλούς τσέχους στρατιώτες στην Ισάφη στο κόσμο. Θέλω να πω σε λεπτομέρειες λοιπόν για όλα αυτά στο κείμενο, αλλά θα ήθελα να βρω μια κοινή λύση, μια κοινή διατύπωση με τον Έρμαρ Μπρόκ και τον ε, α, κύριο Ντάφ για να ενθαρρύνουμε με τον σωστό τρόπο το τσεχικό κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συνθήκη της Λισαβόνας για να ενισχυθούν οι εξουσίες του Τσεχικού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Θα καταθέσω τι δικέ μου τροπολογίε, αλλά να θυμηθείτε ότι δεν είμαστε Ιρλανδία. Είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πετύχει πολλά πράγματα και ελπίζω θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ κυρία Χιμπάσκοβα. Κατάλαβα τι εννοείτε. Επειδή την Παρασκευή θα είμαι στην Πράγα θα κάνω ό,τι μπορώ. Ο κύριος Γιούρι, τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση <clears throat> με την γνωμοδότηση του κυρίου Νταφ, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα που συνδέεται με το σημείο 10. Αυτό που λέμε εδώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αξιολόγηση των ε, κοινοβουλευτικών βημάτων και έχουμε τρία τέτοια βήματα κατά περιοχή. Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί στο Εθνικό Κοινοβούλιο όπου μετήχα της χώρας μου ήμουνα μέλος της συνέλευσης της Ευρωμεσογειακής και είχα παρακολουθήσει το έργο αυτής της συνέλευσης. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας αυτών των βημάτων, αυτών των φόρα, χωρίς να έχουμε εταίρους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε σε επαφή. Μπορούμε να δώσουμε μονάχα την οπτική γωνία της Ευρώπης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση, εκτός αν και οι εταίροι μας είναι έτοιμοι να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Δεν θέλω λοιπόν αυτά τα κοινοβουλευτικά φόρα να φαίνονται ότι είναι περιτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντάφ, αν έχετε σχόλια. Νομίζω ότι έχω και είμαι ευγνώμων σε όσους μίλησαν. Κυρίως τη δήλωση από τσέχους βουλευτές ότι θα έχουμε μια γρήγορη και επιτυχή περάτωση αυτής της ε, παρατεταμένης και σχετικά επώδυνης διαδικασίας της ε, κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Σαφώς, επειδή έχω πάει στην Πράγα, μάλιστα πάρα πολλές φορές τώρα τελευταία, Είμαι και το, έχω πάει και την τωρινή περίοδο και το φθινόπωρο πολλές φορές και καταλαβαίνω πολύ καλά τις αποχρώσεις που χρησιμοποιούν τα ε, τσέχικα κόμματα στην πολιτική για να μπορέσουν να δουν τι γίνεται με αυτό το διαλυφωλονικούμενο ζήτημα στην Πράγα. Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα που θέσατε, το θέμα της χρηματοδότησης, υπάρχει μια διάκριση στη συνθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ σαφής για το κοινό κόστος ε, της ΚΕΠΑ και της ε, ΚΕΠΑ τα οποία θα βαρύνουν εμά από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βαρύνουν και εμάς ως ε, κοινή αρχή προπολογισμού. Δεν ξέρω βέβαια ως ε, προς την έκταση και το χρονοδιάγραμμα της ε, χρηματοδότησης της ΚΕΠΑ και των επιχειρήσεών της. Και ως προς την ταχύτητα με την οποία θα αυξηθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό πρόκειται για ένα ε, πολύ σημαντικό στοιχείο του τι θα γίνει αυτή τη στιγμή ξεκινήσει η διαδικασία πολύ σύντομα μετά από την θέση εφαρμογή της συνθήκης. Εκείνο επίσης που είναι σαφές είναι ότι το κόστος των επιτόπου επιχειρήσεων ως προς τα στρατεύματα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η πάγια λύση του προβλήματος, αλλά θα είναι μία λύση ή μάλλον η άγουσα που θα ακολουθήσουμε βάσει της συνθήκης που προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή. Συμφωνώ ότι στόχος μας είναι το Συμβούλιο. Η κυρία Ονρόιτε έχει δίκιο. Θα πρέπει όλοι από κοινού να εστιάσουμε στους υπουργούς. Μπορούμε συλλογικά να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε αυτή την κατάσταση, όντας ενημερωμένοι, όντας παρόντας ε, και πολύ δραστήριοι ε, να ελέγχουμε τα, συνεχώς τι ακριβώς συμβαίνει. Ως προς την Κόζακ, πολύ σωστό το ερώτημα που θέσατε. Είναι σημαντική και θα καταφέρει να ευμερίσει. Νομίζω ναι, αλλά η λειτουργία της θα πρέπει να θεωρείται περιορισμένη. Είναι υπόκειται στον έλεγχο και των Εθνικών Κοινοβουλίων και των δικών μας. Ως προς την ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα πράγματα τα οποία έχουν αποτέλεσμα και αυτά τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα και την διαφορά στην προσέγγιση μεταξύ 27 Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συχνά υπάρχουν και διαφορές μεταξύ άνω και κάτω βουλής του ίδιου του Εθνικού Κοινοβουλίου. Έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές πρακτικές ε, ε, και διαφορετική νοοτροπία ως προς τον ε, έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της πολιτικής εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ε, εξαγάγουμε συμπεράσματα από αυτή την κοινή αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιημένη εμπειρία ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε και σαφώς θα πιστεύω ότι θα μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει ίσως να ε, μεταλαμπαδεύσουμε όλες αυτές τις γνώσεις λίγο περισσότερο από όσο τις ε, διαδίδουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό μήνυμα από την Κόζακ και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Στην έκθεση Μπροκ για την ΑΦΚΟ προτείνονται κάποια πράγματα για την αύξηση της παρουσίας και της συμμετοχής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός των Εθνικών Κοινοβουλίων και πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε η εμπειρία της Άνω Βουλή τη Ολλανδία που φαίνεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα, Επομένω θα μπορούσαμε και, εμείς να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη από αυτή την εμπειρία. Τέλος, η πρότασή μου στην παράγραφο 10 να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτών των φόρα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να θέσουμε στην ημερήσια διάταξη των κοινών ε, συνεδριάσεων που κάνουμε τρεις φορές ε, το χρόνο. Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε για την άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων από αυτόν. Ποια είναι η δική τους η πείρα. Πιστεύω ότι θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων να δούμε ακριβώς για ποιον είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα και για ποιον έχουν αποτελέσματα ή για ποιον δεν έχουν. Και αυτό θα υποχρέωνε τη δική μας την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων να είναι προετοιμασμένη για μια τέτοια συζήτηση. κάνοντας μια εσωτερική αξιολόγηση, την οποία πιστεύω ότι όλοι θα βρούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Κύριε Νταφ, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 16 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Έλεγχος του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα προενταξιακά μέσα είναι τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Βλέπω ότι η κυρία Κράτσα είναι παρούσα και ο συντάκτη γνωμοδότηση είναι ο συνάδελφο Ιστβάν Σεντ Ιβάνι. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να τονίσω μόνο τα κύρια σημεία του σχεδίου και μετά μπορείτε να συζητήσετε από τη στιγμή που θα υπάρχει το σχέδιο σε έγγραφη μορφή. Το πρώτο και πιο σημαντικό σημείο είναι η ανάγκη να δώσουμε σε όλες τις χώρες που είναι αποδέκτριες πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία πολιτικής. Αυτό είναι το βασικό θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί. Και επίσης ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στις περιοχές που δίνουν άμεσο όφελος στους πολίτες. Να δείξουμε ότι όλα αυτά γίνονται για τους ίδιους τους πολίτες και προς το δικό τους τελικό όφελος. Τρίτον, λυπούμεθα που τα πρώτα προγράμματα είπα ενεκρίθησαν μονάχα στο τέλος του 2007 και μερικά από αυτά το 2008. Επομένως, ως εκ τούτου δεν έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο για να κρίνουμε για την εφαρμογή τους και τον τρόπο λειτουργία τους. Θέλω λοιπόν να παρακινήσω την Κομισιόν να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό στην εφαρμογή των σχεδίων αυτών και να δώσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για όλα αυτά. και θα πρέπει να πιέσουμε την Κομισιόν να αυξήσει τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα για τους νέους, το Erasmus Mundus, το Tempus κτλ. Και χαιρόμαστε για την εμπλοκή πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς αυτούς. Θα θέλαμε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για τη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος προξενικών θεωρήσεων, όπως αναφέρεται στο οδικό χάρτη και οι, τα προγράμματα ΙΠΑ μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτά. Εγώ δεν έχω προβλήματα με τις τροπολογίες, αλλά έχετε τώρα κάποια ερωτήματα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Λέει στα Ουγγρικά ο κύριος Γκάλερ. Η κυρία Κράτσα ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας αυτή την σύντομη συζήτηση που γίνεται ε, για την ε, γνωμοδότηση του πρωτοξιακού μέσου στην ε, <clears throat> που εγίνεται σήμερα και ήθελα να σας πω ότι συμμερίζομαι τον εισηγητή σας για την καθυστέρηση έγκρισης και όπως τονίζω και εγώ στην έκθεση ε, <clears throat> είναι πολύ σημαντικό και, και οι δύο επιτροπές, τόσο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσο και η δική μας ελέγχου του προπολογισμού, να επιστήσουν την προσοχή και της Επιτροπής και του Συμβουλίου στο σημείο αυτό ακριβώς ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουν ε, οι χρηματοδοτήσεις και να, η, η καθυστέρηση αυτή που έγινε να αποτελέσει άλοθη για τη διακοπή της φυσιολογικής ε, ε ροής ε, χρημάτων και προγραμματισμού προς τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες. Επίσης ένα άλλο ε, σημαντικό θέμα το οποίο τονίζουμε και πιστεύω ότι συμμερίζεστε είναι ότι τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων ΦΑΡ, ΣΑΠΑΡ, ΙΣΠΑ σε χώρες ε, μέλη σήμερα ε, ε, υποψήφιες παλιότερα πρέπει να προσέξουμε να μην επαναληφθούν. Αυτό είναι και αν θέλετε και το κίνητρο της έκθεσης πρωτοβουλίας που κάνει η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών να αποτελέσει έστω αυτή την πρώιμη φάση εφαρμογής να αποτελέσει ένα κίνητρο για παρακολούθηση και προσοχή και γι' αυτό ζητούμε και ε, από το ελεκτικό συνέδριο να εκπονήσει μια ειδική έκθεση ενδιάμεση αξιολόγησης και ε, εφαρμογής του προνοτοξιακού μέσου. Επίσης κάτι άλλο που ε, η έκθεση η δική μας τονίζει είναι από τα συμπεράσματα, αυτά τα ε, προκαταρτικά συμπεράσματα που έχουμε μέχρι σήμερα, πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να ευθεγραμμίσει καλύτερα το ενταξιωτικό μέσο σε κάποιους τομούς και στόχους της προτεραιότητας των εκθέσεων πρόοδου και ενδεικτικά να φέρουμε το περιβάλλον, το διαπολιτισμικό διάλογο, τα δικαιώματα των γυναικών, τα κοινωνικά φαινόμενα όπως την ανεργία, τη διασυνοριακή και διακοινωτική συνεργασία, την ασφάλεια, την πυρονική. Είναι ένα θέμα της ε, της ε, περιοχής. Εμείς θα συζητήσουμε την έκθεση στις 17 Φεβρουαρίου και ο εισηγητής της νομοδότησης, όπως και τα άλλα μέλη που ενδιαφέρονται, ε, είναι καλοδεχούμενα στην Επιτροπή μας για να έχουμε μια ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί η Θα δίνω το λόγο στην Κομισιόν αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Εάν θέλετε, πάντα. Ευχαριστώ. Καταγράψαμε με ενδιαφέρον την έκθεση του εισηγητού. Συμφωνούμε με τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίδει η έκθεση και θα παράσουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνει η Επιτροπή για να ε, αντιμετωπίσει τα ζητήματα στην βάση αυτή των γραμμών στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε Σέντιβάνη, ούτε κι εσείς. Έχει κλείσει λοιπόν το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και έχουμε το επόμενο σημείο. Δημοσιονομικές πτυχές της μεταρρυθμιστικής συνθήκης. Επί της ουσίας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών Αρμόδια και ο συντάκτης νομοδότησης είναι και πάλι ο συνάδελφος του Σεντ Ιβάνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε τα ουγγρικά σας βελτιώνονται από στιγμή σε στιγμή. Και τώρα θα είμαι σύντομος και θα είμαι, διότι η προηγούμενη συζήτηση για την έκθεση DAF ασχολήθηκε με πολλά από τα θέματα που θα συζητήσουμε τώρα. Πρώτον, συζητήσαμε πολλές φορές τη συνθήκη της Λισαβόνας και ξέρουμε ότι θα έχει και κάποιες οικονομικές ουσιαστικές πτυχές στην εξωτερική πολιτική. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Δεν είμαστε σε θέση τώρα να καταλήξουμε σε τελικές δημοσιονομικές εκτιμήσεις, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, καταρχάς, ενώ ελπίζουμε και προσδοκούμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υπάρχει σαφές πρόγραμμα αντιμετώπισης των μέτρων εξορθολογισμού, διότι περιμένουμε ουσιαστική μείωση του διοικητικού κόστους. Τέλος πάντων, με όλα αυτά σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική εικόνα, τελική εικόνα των οικονομικών διαστάσεων. Το θεσμικό ε, πλαίσιο είναι βέβαιο. Η Δημοσιονομικές λοιπόν δεσμεύσεις θα πρέπει να γίνονται σταδιακά όπως καθώς δημιουργούνται τα διάφορα θεσμικά όργανα. Αυτό σημαίνει δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα νούμερα. Λόγω τη της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης τονίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πίεση στις κατηγορίες 4 και 5. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Για την... Στο μέτρο που η επερχόμενη δημοσιονομική εξέταση παρέχει περαιτέρω πόρους στην κατηγορία 5, θα πρέπει να ζητήσουμε σημαντική αύξηση και πραγματική αύξηση των MFF. Θα το συζητήσουμε αύριο αυτό. Και προφανώς μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση του νέου θεσμικού πλαισίου. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Για τη Λισαβόνα, όπως ξέρετε, δημιουργούνται νέες διαδικασίες ευπρόσδεκτες που θα επιτρέπουν ταχεία πρόσβαση στον προπολογισμό της Ένωσης, κάτι σημαντικό. Πρέπει να πω εδώ ότι κατά την άποψή μου κάθε εξωτερική δράση θα πρέπει να να χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδυλία και μόνο κατε, σε επίουσες περιπτώσεις από τα κράτη-μέλη. από εισφορές δηλαδή ad hoc εισφορές των κρατών μελών. Για την εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών ζητούμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν έγκαιρα συγκεκριμένη εικόνα των θεσμικών ρυθμίσεων και των συναφών οικονομικών υποχρεώσεων, τόσο ώστε να έχουμε ένα ουσιαστικό, βιώσιμο, τελικό πλάνο. Κύριε Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαιρετίζει το σχέδιο του κυρίου Σεντιβανή. Εμείς καταγράφουμε τα σχόλια, μάλλον το, το περιεχόμενο των σχολείων του κυρίου Σεντιβανή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα η Κομισιόν. Μπορούμε να πω ότι ήδη στα έγγραφά μας για το προϋπολογισμό που τα οποία είναι δημόσια έχουμε καταγράψει ότι μπορεί η θέση εφαρμογή τη συνθήκη να έχει επιπτώσει επί του προπολογισμού και θα επανέλθουμε εν καιρό στη διαδικασία του προπολογισμού. Σύμφωνα με τον κύριο Σφεντιβάνη είναι πολύ νωρί για να έχουμε συγκεκριμένε εκτιμήσει των συνεπειών του προπολογισμού εάν κάτι τέτοιο προκύψει και για την Κομισιόν είναι πάρα πολύ πρόωρο να πούμε τι συνέπειες θα προκύψουν και κατά πόσον αν το κάνουμε τώρα θα προκαταλάβουμε κατά κάποιο τρόπο αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν εν καιρό εάν και όταν εγκριθεί η συνδίκη της Λισαβόνας. Τεθεί σε εφαρμογή συνδίκη Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο από τους συναδέλφους. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς σα ανακοινώνω ότι λόγω του περιθωρίου τροπολογιών είναι στενό το περιθώριο αυτό 19 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα και λόγω της στενότητας χρόνου σας παρακαλώ εξαιρετικώς να καταθέσετε τροπολογίες στα αγγλικά και μόνο. Αυτή ήταν η μέρη διαταξία σήμερα. Σας ευχαριστώ. Και αύριο πουρνό πουνό στις 9 συνεχίσουμε.